Σας ευχαριστούμε κύριε υποψήφια επίτροπε για την εισαγωγική σας αυτή παρουσίαση και χωρίς άλλη χρονοτριβή θα περάσουμε στη διαδικασία των ερωταπαντήσεων. Πρώτη ομιλήτρια θα είναι η κυρία Μαγκίνες από το ΕΛΚ. Παρακαλώ κυρία Μαγκίνες υποβάλλετε την ερώτησή σας και επαναλαμβάνω χρόνου φίδου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Επίτροπο. Στα πλαίσια της εισαγωγής σας αναφερθήκατε στην γεωργική παραγωγή και τις αγορές. Το τέλος όμως της τροφιμικής αλυσίδας είναι ο τομέας του λιανικού εμπορίου. Εκεί έχουν προβλήματα σε σχέση με, την, με τον τομέα αυτό και οι γεωργοί. Ε, σαν παράδειγμα η διαδικασία την οποία, με την οποία με διαγωνισμούς προμηθεύεται προϊόντα οποροκυπευτικά η αλυσίδα Aldi καταστρέφει τον τομέα αυτό στην χώρα μας. Λοιπόν, ε, είχε πάρει κάποιες δράσεις, είχε αναλάβει κάποιες δράσεις η προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι θα κάνετε εσείς σαν υποψήφιος ε, επίτροπος ε, για να ε, δώσετε μια απάντηση και να βγάλετε το φόβο από τους γεωργούς. Εξαρτάται το, τα έσοδα των γεωργών εξαρτώνται από αυτές τις διαδικασίες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η υπερσυγκέντρωση του λιανικού τομέα την τελευταία δεκαετία έχει οδηγήσει σε μια ανισότητα θα έλεγα σε σχέση με το διαπραγματευτικό πλαίσιο και γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποιες ε, συμβατικές σχέσεις όπως επίσης ε, και κάποιες διαπραγματευτικές πρακτικές των ισχυρών στον τομέα αυτό με διαφορετικό τρόπο. Αυτές οι στρεβλές πρακτικές οι εμπορικές πρέπει ε, να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο. Δεν έχουμε όμως ίσως το κατάλληλο πλαίσιο γι' αυτό. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες για αντίδραση από πλευρά των γεωργών. Συνεπώς, εγώ θεωρώ ότι η πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει τρόπους εφαρμογής της νομοθεσίας στα κράτη-μέλη και έχουμε το τελευταίο παράδειγμα της ε, Ιρλανδίας ε, για να αντιμετωπιστούν αυτές οι στρεβλές πρακτικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι έτοιμη να προτείνει και νομικά μέσα εάν το διοικητικό επίπεδο και οι διαπραγματεύσεις δεν λύνουν τα προβλήματα αυτά, κάτι το οποίο φαίνεται ότι δυστυχώς συμβαίνει. Και αυτά θα τα συζητήσω με σας εφόσον με επιλέξετε, έτσι ώστε να πετύχουμε μια δίκαιη τιμή για τον παραγωγό και όχι την ελάχιστη τιμή που έχουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Δεκάστρο. Έχετε το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, η πρόταση όταν μας παρουσιάστηκε για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ υπήρξαν συνάδελφοι που είπαν ότι είναι ένα εμπόδιο ουσιαστικά, ένα βάρος για τους γεωργούς. Προσπαθήσαμε να την βελτιώσουμε, να μετριάσουμε τις επιπτώσεις, αλλά όχι απολύτως. Στην ουσία θα έπρεπε να τονίσουμε την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τη θέση των προϊόντων μας στις διεθνείς αγορές. Ε, θα μπορέσετε εσείς να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες που δίνει η μεσοπρόθεσμη ε, αναθεώρηση για να βελτιώσετε την κατάσταση. Ε, επίσης ε, φαίνεται ότι κάποιοι λένε ότι εσείς δεν είσαστε υπέρ του διαλόγου και προτιμάτε να δράτε φυσικά με μέσα τα οποία δεν είναι απολύτως ε, ε, σωστά επικοινωνιακά. Well, first of all, can I say... Καταρχάς, φυσικά θα συνεργαστώ πλήρως με την Επιτροπή σας και το Κοινοβούλιο κατά την άσκηση των καθηκόντων μου Επιτρόπου. Βεβαίως μπορεί να υπάρξουν εξαιρετικές καταστάσεις, αλλά θα είναι εξαιρέσεις. Αλλά δεσμεύομαι σήμερα στην εισαγωγική μου ομιλία, να συνεργαστώ στενά με την Επιτροπή σας, να κάνω πάντα, να λογοδοτώ πάντα, να είμαι πάντα ε, διαφανής και προσβλέπω στις επίσημες και ανεπίσημες επαφές με την Επιτροπή σας για να προωθήσουμε τους στόχους μας. Σίγουρα δεν θα θεωρήσω ότι είναι ανεπαρκής η συνεργασία μου με τους συναδέλφους πολιτικούς για την αναθεώρηση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Είμαι πεισμένος ότι η νέα ΚΓΠ είναι ουσιοδός πιο πράσινη από την προηγούμενη. Για πρώτη φορά 30% των αμέσων πληρωμών είναι υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν ε, συμπληρωματικές ενέργειες για την ε, ανάπτυξη της υπαίθρου και την προστασία του περιβάλλοντος. Ακούω την ε, τις επικρίσεις ότι η μεγάλη πλειονότητα των γεωργών μπορεί να εξαιρεθούν από αυτό το πρασίνισμα και ένας ουσιώδης αριθμός γεωργών ε, εξαιρούνται εφόσον έχουν κάτω από 15 εκτάρια. Αλλά το 50% της καλλιεργήσιμης γης θα συμπεριληφθεί. Η επίπτωση των ε, μέτρων για το πρασίνισμα που ε, εγκρίναμε στη δήλωση το περασμένο Απρίλιο μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής είναι οπωσδήποτε κάτι το σημαντικό και θα συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη και υπάρχει μια ειδική ενότητα στην Επιτροπή για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη μετά από ένα χρόνο. Λοιπόν, θα εξετάσουμε του τομεί ε, οικολογικού σχεδιασμού ε, και ε, στόχευση. Θα δούμε τι στοιχεία θα έχουμε και βεβαίω δεσμεύομαι να συνεργαστώ πολύ συχνά για τα θέματα αυτά με τα μέλη του Κοινοβουλίου και τα κράτη-μέλη. Πολύ καιρό χρειάστηκε για να φτάσουμε σε αυτή την πολιτική. Ξέρω ότι το Κοινοβούλιο ε, συμμετείχε πολύ σε αυτή τη διαδικασία, πολλές τροπολογίες που υποβάλλεται στην αρχική πρόταση. Θα δούμε λοιπόν μετά από ένα χρόνο πώς θα έχουν λειτουργήσει τα πράγματα στην πράξη. Σας ευχαριστώ, ο κύριος Νίκολσον. Κύριε Επίτροπε, κύριε υποψήφια Επίτροπε, όταν έγιναν μέλος της Επιτροπής, το 1999 η κοινή γεωργική πολιτική ήταν γύρω στο 55% του προπολογισμού. Τώρα είναι λιγότερο από 40%. Τότε είχαμε ε, τα βουνά γάλακτος, τα βουνά βοήου κρέατος. Τώρα όμως ε, στην ουσία είμαστε καθαροί εισαγωγή για τα προϊόντα αυτά. Όλοι μιλάνε για επισητιστική ασφάλεια. Κατά την ε, αναθεώρηση της ΚΑΠΑΓΑΜΑΠΗ δεν έγινε τίποτα για να τη διασφαλίσει. Τώρα έχουμε υπερβολική ε, γραφειοκρατία και διαδικασίες και δεν έχει υπάρξει απλούστευση. Θα κάνετε ό,τι μπορείτε ούτως ώστε η Γεωργία να είναι και πάλι η πρώτη προτεραιότητα των επιτρόπων. Θα υπερασπιστείτε οποιασδήποτε, θα αντιτεθείτε σε οποιασδήποτε περαιτέρω περικοπές και θα κάνετε ό,τι μπορείτε ούτως ώστε η καινή γεωργική πολιτική να βοηθάει τους γεωργούς. Ξέρετε τώρα που θα λήξουν οι ποσοστώσεις τον επόμενο Μάρτιο. Έχετε δυνατότητα να αντιδράσετε ούτως ώστε οι παραγωγοί γαλακτοκομικών να έχουν επαρκές επίπεδο ε, ε, παρέμβασης και πρόσβαση στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων. Ο κύριος Χόγκαν. Φυσικά θα επερασπιστώ όσο μπορώ τον προπολογισμό, αλλά φυσικά ο ρόλος του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είναι πολύ σημαντικός για τον προπολογισμό. Έχουν γίνει προτάσεις και εσείς θα συμβάλλετε βεβαίως ε, στεναρά θα προτείνετε, ε, θα έχετε αντιρρήσεις αν υπάρξει ε, προσπάθεια περικοπής του γεωργικού προπολογισμού. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να επαγρυπνούμε. Θα συνεργαστώ επίσης πολύ στενά με τον Επίτροπο για τον προπολογισμό, ούτως ώστε ο προπολογισμό για τη γεωργία να είναι δίκαιος. Συμφωνώ με αυτά που είπατε ότι υπάρχει ανησυχία για τη γραφειοκρατική φύση κάποιων μεταρρυθμίσεων. Δεσμεύομαι ότι θα, θα μειωθεί η γραφειοκρατία και θα υπάρξει απλούστευση την επόμενη πενταετία και φυσικά ήδη θα ξεκινήσω τον έλεγχο, το screening των διαφόρων μέτρων στο γεωργικό τομέα, να δούμε τι μπορούμε να απλουστεύσουμε και θα συνεργαστώ με τον πρώτο αντιπρόεδρο Τίμερμανς για να ε, το επιτύχουμε. Τα πρόσφατα γεγονότα σε σχέση με την κρίση Ρωσίας-Ουκρανίας φυσικά σημαίνουν ότι χρειαζόμαστε ένα δίχτυο ασφαλείας στον τομέα αυτό. Αυτά που είπατε για το γάλα, αλλά και για άλλα προϊόντα, είναι ε, απόλυτα δικαιολογημένα. Αλλά έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδο από την μεταρρύθμιση Μαξάρ 92 και μετά, το ώστε η πολιτική μα να έχει προσανατολισμό προ την αγορά, έχει λειτουργήσει. Οι τιμέ ε, στην παγκόσμια αγορά και οι δικέ μα τιμέ έχουν προσεγγίσει πολύ. Θα μπορούσαν να προσεγγίσουν περαιτέρω. Θεωρώ λοιπόν ότι οι καταργήσεις των περιορισμών ε, ε, της παραγωγής στο γάλα και στη ζάχαρη είναι μια ευκαιρία για περισσότερη αγορά, περισσότερες ε, θέσεις εργασίας και οι προτάσεις που θα κάνω τα επόμενα χρόνια είναι ότι πρέπει να διαφοροποιήσουμε την διάθεση των προϊόντων μας από περιοχές που είναι ευαίσθητες για να έχουμε περισσότερες δυνατότητες διάθεσης των προϊόντων μας σε άλλες αγορές. Και δεσμεύομαι να δώσω το καλό παράδειγμα και σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρόντε. Καλημέρα σας κύριε Χόγκαν. Χαιρόμαστε που σας ξαναβλέπουμε. Και μου άρεσαν πολύ αυτά που είπατε στην εισαγωγική σας παρουσίαση. Χαίρομαι που είπατε ότι δεν είναι και πολύ απλά όλα αυτά τα πράγματα. Μία από τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί μας και μάλιστα καθημερινά είναι η άνηση εφαρμογή μιας ε, σειράς κανονισμών και οδηγιών στα κρατημέλη. Αυτή η άνηση εφαρμογή δημιουργεί άδικο και αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ των γεωργών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει να επισημάνουμε ότι χωρίς καλό ανταγωνισμό και ίσες συνθήκες ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίσουμε χαλεπούς καιρούς όταν ξεκινήσουμε εμπορικές συμφωνίες με άλλες χώρες με τρίτες χώρες. Πώς θα εξασφαλίσετε λοιπόν ε, ε, δίκαιο και θεμητό ανταγωνισμό στη Γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί γνωρίζουμε ότι το screening, ο διεξοδικός έλεγχος και τα στενά χρονοδιαγράμματα δεν πρόκειται να επιτύχουν το στόχο μας. Σας ευχαριστώ. Το 2016 η Ευρωπαϊκή Ένωση για πρώτη φορά έγινε ε, αμυγής εξαγωγέας τροφίμων. Και το 2013 ξαναγίναμε ε, αμυγής εξαγωγές, γιατί στο διάμεσο διάστημα είχαμε αύξηση και των εισαγωγών. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό το θέμα να έχουμε μια γεωργία που θα είναι στραμμένη προς την αγορά. Το είπα αυτό και προηγουμένως, αλλά και στην εισαγωγική μου ομιλία. Και θα πρωτοστατήσω στις εμπορικές ε, συμφωνίες προκειμένου να δημιουργηθούν εμπορικές ευκαιρίες ε, για τους γεωργούς μας σε άλλες χώρες. Βέβαια, για να στεφθεί με επιτυχία η ανταγωνιστικότητά μας, θα πρέπει να επιτρέψουμε με τις μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ που θα είναι στραμμένες προς την αγορά να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα, να έχουμε πιο αποτελεσματική γεωργία και να έχουμε και αποτελεσματικό ανταγωνισμό. Θα ενισχύουμε τις οργανώσεις παραγωγών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε όλο και μεγαλύτερη συγκέντρωση ε, κατάντη στην αρχή της ε, αλυσίδας τροφίμων μεταξύ των παραγωγών, ιδιαίτερα στα προκυπευτικά και στο γαλακτοκομικό τομέα. Οπότε η, η μείωση της γραφειοκρατίας, ο περιορισμός του γραφειοκρατικού άχθους και μία πολιτική που θα είναι στραμμένη στην αγορά θα είναι οι βασικές αρχές που θα ε, χαρακτηρίσουν την πολιτική μου την επόμενη πενταετία. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σένερα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα πορτογαλικά. Η ευρωπαϊκή πολιτική της για τη Γεωργία ε, καταστρέφει κάθε μέρα χιλιάδες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Θέλετε μια νέα ΚΑΠ που θα εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές εισόδημα στα, στους γεωργούς που θα εξασφαλίζει την ευημερία των ε, ζώων. Μια νέα ΚΑΠ που θα βελτιώνει την κατανομή των άμεσων ενισχύσεων. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να θεσπιστούν κάποια μέτρα για να αποφευχθούν κρίσεις σαν αυτές που θα δημιουργηθούν στο γαλακτοκομικό τομέα με την κατάργηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων. Ποια μέτρα θα προτείνετε για την αγορά. Μιλήσατε για το TTIP εγώ θα μπορούσα να μιλήσω για το ΣΕΤΑ, τη συμφωνία δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά. Σε ποιους γεωργικούς τομείς θα εφαρμοστούν οι συμφωνίες αυτές και τι θα κάνετε προκειμένου να υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις προτάσεις σας. Νομίζω ότι οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν τεθεί σε εφαρμογή δείχνουν το αντίθετο από αυτά τα οποία είπατε. Έχουμε ένα βασικό εισόδημα για τους γεωργούς στην Ευρώπη πλέον. Έχουμε μέτρα για το λεγόμενο πρασίνισμα οικολογική διαχείριση, το οποίο προσφέρει και αυτό κάποια εισοδήματα. Για κάποια μέτρα για τους μικρούς γεωργούς ε, έχουν υπάρξει συγκεκριμένες προβλέψεις μέχρι 5.000 ευρώ και ιδιαίτερα για αυτούς που έχουν ε, λιγότερο από 5 εκτάρια. Υπάρχει λοιπόν μια πρόκληση έτσι ώστε να υπάρξει ένας βιώσιμος γεωργικός τομέας που θα παράγει τα προϊόντα που χρειαζόμαστε το βάρος που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι γεωργοί πρέπει φυσικά να αντιμετωπιστεί και εν μέρει έχει αντιμετωπιστεί και μέσω του πρασινίσματος και μέσω των στοχευμένων μέτρων για οικολογικού ενδιαφέροντος περιοχές οι κάτω των 5 εκταρίων έχουν εξαιρεθεί και υπάρχουν φυσικά και περαιτέρω στηρίξεις μέσω της αναδιανομής των πόρων έχουν γίνει λοιπόν προσπάθειες και από την προηγούμενη Επιτροπή κατά τη διάρκεια της τελευταίας κοινοβουλευτικής περίοδου για να στηριχθούν τα εισοδήματα των γεωργικών οικογενειών για τη γαλακτοπαραγωγή. Υπήρξαν κάποιες αποφάσεις από το 2008 και μετά οι κανόνες ισχύουν, έχουν υπάρξει αυξήσεις κατά 1%, ε, κάτι το οποίο δείχνει ότι λειτουργήσαν οι τελευταίες προτάσεις. Δεν θα ήταν σωστό να αλλάξουμε τους κανόνες. Ο κόσμος έχει, οι παραγωγοί έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους και ήδη από τον επόμενο χρόνο θα εξετάσουμε την κατάσταση της γαλακτοπαραγωγής. Νομίζω ότι 20 χώρες δεν εξάντλησαν τις ποσοστώσεις τις οποίες είχαν στη διάθεσή τους έτσι και αλλιώς. Ευχαριστώ. Κύριο Χόισλινγκ. Äh, ως Ιρλανδός ήσασταν ε, υπεύθυνο για το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες οδηγίες έγιναν πολύ πιο αδύναμες το οποίο είχε ως επίπτωση να ε, υπάρξουν προβλήματα με την ποιότητα του ποσίμου ύδατος. Θα είστε λοιπόν, ε, θα επαγρυπνήσετε ποτέ για να μην υπάρξουν τέτοια προβλήματα. Θα επαγρυπνήσετε ως Επίτροπος. Επίσης ε, θα είναι η απλούστευση κέντρο βάρους της εργασίας σας. Φυσικά η γεωργική δραστηριότητα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Πρέπει να μειωθούν αυτές. Τι θα κάνετε για τα βιολογικά προϊόντα. Δεν είπατε τίποτα για την βιολογική γεωργία. Τι θα κάνετε για να την προωθήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε εισαγάγει μια σειρά από συμπληρωματικά μέτρα τα οποία είναι φιλικά προς το περιβάλλον και στην Ιρλανδία. Έχουμε λοιπόν πολλά συμπληρωματικά ε, μέτρα και αυτά είναι υποχρεώσεις φυσικά βοηθούν τους γεωργούς και ορισμένοι έχουν τα αντίστροφα παράπονα από αυτά που είπατε. Έχετε δίκιο όμως, δύο κράτη-μέλη ζήτησαν να ληφθούν ειδικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν την πολύ δύσκολη κατάσταση. Τους δόθηκε αυτή η δυνατότητα. Είναι που έχει επιπτώσεις γεωργούς, αλλά η αρχή της ε, συνυπευθυνότητας ε, είναι κάτι το οποίο το διαχειρίζεται το, η οδηγία η οδηγία για να έχουμε καλή ποιότητα υδάτων και επίσης πρέπει να εφαρμόσουμε άλλα μέτρα για το πρασίνισμα όπου καταφέραμε να ε, ε, εφαρμόσουμε τις οδηγίες για τα νητρικά άλατα. Οπωσδήποτε θέλουμε να προστατεύσουμε τους ε, φυσικούς μας πόρους, το νερό. Πέρασα 3,5 χρόνια ε, στην Ιρλανδία για να πίσω τον πληθυσμό να καταλάβει την αξία της καλής ποιότητας νερού, ε, να εφαρμόσουμε την αρχή του ομολύνων πληρώνει και να έχουμε το σωστό, τη σωστή ποιότητα ύδατος. Για τα βιολογικά προϊόντα, ξέρω ότι είστε εισηγητής για μια πρόταση για την βιολογική γεωργία και ε, προσβλέπω στη συνεργασία. Φυσικά δεν πρέπει να καθυστερήσει αυτή η πρόταση. Θα πρέπει να επιταχυνθεί η εξέτασή της ε, μέσα από το Κοινοβούλιο και παρακαλώ τα μέλη της Επιτροπής να μας επιτρέψουν να ε, περάσει με μια απλοποιημένη διαδικασία γιατί πιστεύω ότι μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξη σε πολλά κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Άγγινου. Καλημέρα σας τα κακά μαντάτα είναι ότι θα έχετε δύο κράσει σήμερα. Θα δεχτείτε από την εκλογική μου περιφέρεια πρόκληση ώστε να μπορέσετε να δώσετε ε, μερικές εξηγήσεις για να ακούσετε τις ε, γνώμες των βαβακοπαραγωγών και, τις, ε, και να έρθετε και στην ε, δική μου φάρμα ε, που δείχνει πραγματικά πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις μέλισσες. Επίσης, ε, να επισκεφτείτε κάποιες ε, κτηνοτροφικές ε, φάρμες για να δείτε πώς είναι οι κτηνοτρόφοι που έχουν ελεύθερη βοσκή στα ζώα τους. Επίσης να δείτε πόσο περιοριστικός είναι ο κανονισμός για τα φυτοφάρμακα και να δείτε πόσο δύσκολα είναι να εφαρμόσουμε όλους τους ε, κανονισμούς για την ε, γεωργία και τα φυτοφάρμακα. Ελάτε, σας προσκαλούμε. Ανοιχτή πρόσκληση. Well, don't Κοιτάξτε, μην περιμένετε να, να είμαι και εργατικό χέρια για την ε, εκμετάλλευσή σας. Καλύψατε πάρα πολλά θέματα. Ε, δεν τα ξέρω αυτά που είπατε και για τις ε, μέλισσες και για την βιοπικιλότητα ε, είναι θέματα τα οποία ίσως και εσείς δεν φροντίζετε πολύ γιατί ξοδεύετε εδώ περισσότερο το χρόνο σας. Πάντως θα επισκεφθώ πολλές περιοχές και ελπίζω να μπορέσω να επισκεφθώ και τη δική σας χώρα ε, κατά τη διάρκεια της επόμενης πενταετίας παρά τις δυσκολίες και τις διαφορές που μπορεί να έχουμε. Γνωρίζω ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε γεωργική εκμετάλλευση. Και εσείς και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής σας έχετε ορίσει τον τρόπο που θα εξελιχθεί η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ τα επόμενα πέντε χρόνια. Ας συνεργαστούμε λοιπόν για να μπορέσουμε να σεβαστούμε τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει σχετικά με την εναρμόνιση των κανόνων κτλ. Θα επισκεφθώ ε, κάποια αγροκτήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ίσως και το δικό σας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ήταν καλό να ακούμε λίγο κάτι το διαφορετικό και μετά να γελάμε και λίγο. Η κυρία Ντότζ. Ευχαριστώ κύριε υποψήφια. Σας καλωσορίζουμε εδώ. Ο γαλακτοκομικός τομέας και σημείωσα αυτά τα οποία είπατε βέβαια, αλλά εξακολουθεί να υποφέρει από την πτυτικότητα σε εισαγωγικά των τιμών. Ε, αυτό οφείλεται στο ότι έχει μειωθεί η ζήτηση περισσότερο από όσο προβλέπετο και φυσικά υπήρξε και το εμπάργο για τη Ρωσία. Ε, χτες η προσπάθεια ρύθμισης που έγινε για τις τιμές απέτυχε. Τι θα κάνετε για να προστατεύσετε την γαλακτοβιομηχανία από τις ε, διακυμάνσει αυτές τις τιμές. Και σε ποιο βαθμό μπορεί να προβλέψετε και οι επιστροφές για ε, προϊόντα εξαγωγής ίσως έχουμε αρχίσει να υπερβάλλουμε σε σχέση με το greening, με το πρασίνισμα, με τις οικολογικά στοχευμένες περιοχές. Ε, θα μπορέσετε στα πλαίσια της μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης ε, να βοηθήσετε να γίνουν κάποιες αλλαγές στην γεωργική πολιτική η οποία πράγματι επιβαρύνει προς στιγμήν τους γεωργούς. Αναφυσβήτητα γνωρίζω αυτό το πρόβλημα και είχαμε μείωση κατά 7,3 των τιμών γάλακτος. Είναι ανησυχητικό αυτό στο γαλακτοκομικό εμπόριο, αυτή η φθήνουσα πορεία των τιμών. Και φυσικά το ρωσικό εμπάργο δημιούργησε περαιτέρω προβλήματα. Και αυτή τη στιγμή ε, είχαμε αύξηση της παραγωγής εξαιτία των υψηλών τιμών και της ε, καλοκαιρίας. Και επίση το θέμα ε, της Κίνας και της αύξησης παραγωγής εκεί δεν πρέπει να παραμεληθεί. Πάντως η εργαλειοθήκη που έχουμε με τα μέτρα αγοράς, ε, στα πλαίσια της κοινή οργάνωσης αγοράς, θα αξιοποιηθεί στο, έπαθρο, ε, στο έπακρο, ακόμη και το θέμα των εξαγωγικών επιστροφών. Βέβαια, ε, είναι πολύ δαπανηρός αυτός ο τρόπος προσέγγισης αγοράς, οι εξαγωγικές επιστροφές. Βέβαια, στις κρίσεις χρειάζονται και προστατευτικά μέτρα και θα τα χρησιμοποιήσουμε για να προστατεύσουμε τα εισοδήματα. Θα έχουμε διάμεση επανεξέταση της κοινή αγροτικής πολιτικής, σας το υπόσχομαι, αλλά πρέπει να περάσει ο χρόνος και να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία για να κάνουμε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στο δεύτερο γύρο. Ο κύριος Ντόρφαν είναι ο πρώτος ομιλητής. Äh, Κύριε υποψήφιοι επίτροπε, να συνεχίσω για το γάλα. Παραγωγή γάλακτος στις μειονεκτικές περιοχές, στις ορεινές περιοχές συγκεκριμένα. Πριν από δύο χρόνια κάνετε μια μελέτη για το πώς θα εξελιχθούν οι ποσοστώσεις όταν, και πώς, τι θα γίνει η κατάσταση όταν λήξουν και υπήρχε η αντίληψη ότι όταν καταργηθούν οι ποσοστώσεις θα υπάρχει πολύ μεγάλη συγκέντρωση στην παραγωγή γάλακτο που σημαίνει ότι θα εξαφανιστεί η παραγωγή γάλακτο σε αυτέ τι περιοχέ, τι μειονεκτικές και ορεινέ. Γι' αυτό είχαμε κάνει μια έκθεση πρωτοβουλία όπου προτείναμε μέτρα και ε, θελήσαμε να αντιτεθούμε σε αυτέ τι εξελίξει. Όμω δεν έγινε τίποτα στην πράξη. Σε μερικού μήνε λήγουν οι ποσοστώσει. Υπάρχει κίνδυνο λοιπόν για αυτέ τι ορεινές περιοχέ. Και σε ορισμένε από αυτές τι περιοχές δεν υπάρχει καμία εναλλακτική λύση. Τι μέτρα λοιπόν θα λάβετε τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει σε σχέση με αυτό. Η κατάληξη των διαπραγματεύσεων για την μεταρρύθμιση της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής δίνουν αρκετή ευελιξία στα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να δώσουν ε, εθελοντική βοήθεια. Και 27 από τα 28 κράτη-μέλη θα δώσουν μια τέτοια εθελοντική βοήθεια θα υπάρξει μια ανακατανομή των πληρωμών σε περιοχές που έχουν ε, γεωμορφολογικές ε, αδυναμίες και άλλες δυνατότητες υπάρχουν να στηρίξουμε τους εργαζόμενους, τους γεωργούς στις ε, περιθωριακές περιοχές. Φυσικά η Ήπεθρος και ιδιαίτερα οι πιο ακραίες περιοχές χρειάζονται βοήθεια και πρέπει να δοθεί βοήθεια για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και η κοινωνική συνοχή σε αυτές τις περιοχές. Φυσικά θα το εξετάσουμε αυτό. Πώς εφαρμόζουν λοιπόν τα κράτη-μέλη την ε, μεταρρύθμιση της ΚΚΠ, Να δούμε λοιπόν αν αξιοποιούν και αυτή τη δυνατότητα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει η μεταρρύθμιση της ε, Κουγουπού πριν ε, δούμε τι επιπτώσεις υπάρχουν και σε αυτές τις ακραία περιφερειακές περιοχές. Και υπάρχουν δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιήσουν τα κράτη-μέλη για αυτές τις ακραίες τις πολύ περιθωριακές ορεινές περιοχές. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Αντρίε. Ευχαριστώ. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, εδώ πίσω σας. Οι τρομερές διακυμάνσεις των τιμών ε, δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στη σταθερότητα του εισοδήματο των γεωργών, δημιουργεί κρίσεις και γεωργικές και επισητιστικές. Η πολιτική της απόλυτης φιλελευθερωποίησης των αγορών δεν είναι κατάλληλη για να έχουμε μια ανταγωνιστική γεωργία, μια βιώσιμη γεωργία που να δημιουργεί ανάπτυξη, απασχόληση σε όλες τις περιφέρειες της Ένωσης. Θα κάνετε κάτι για να υπάρξει κάποια ρύθμιση των αγορών, για να διαχειριστούμε τις κρίσεις, να μην επανέλθω στο θέμα του γάλακτος. Ο κύριος Ντόρφμα το ανέφερε μόλις τώρα, ιδιαίτερα για τις ευαίσθητες και ενδιάμεσες περιοχές. Άλλο τομέα. Δεσμεύεστε να γίνει πλήρω σεβαστή η νομοθεσία για, τους, ε, ε, για τις γεωγραφικές ενδείξεις και ιδιαίτερα στις διατλαντικές σχέσεις. Και όσον αφορά ιδιαίτερα τις γεωγραφικές ενδείξεις θα, στον τομέα του ίνου ε, θα κάνετε αυτό που πρέπει, διότι όπως ξέρετε οι Αμερικανοί έχουν τη δυνατότητα να δίνουν ονόματα εκτιμάτων ίνου στο ίντερνετ. Ο κύριος Χόγκαν. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι για τη Γαλλία το θέμα αυτό, γεωγραφικές ενδείξεις. Ονόματα ε, που ε, καταχωρούνται ως ονομασία προέλευσης προστατεύονται πάρα πολύ κατά της απάτης και άλλων καταχρήσεων για προϊόντα που δεν παράγονται εντός της ε, περιοχής που καθορίζει η γεωγραφική ένδειξη, αλλά έχουμε πολλές ενέργειες ως Επιτροπή για να ενισχύσουμε τη δυνατότητα των συστημάτων ελέγχου της Ένωσης κατά των απατών και ιδιαίτερα η Γενική Διεύθυνση ΣΕΝΚΟ έχει ένα δίκτυο ε, εθνικών σημείων επαφής για τα θέματα αυτά, για ανταλλαγή πληροφοριών, για να καταπολεμηθούν οι απάτες. Ιδίως αν είναι διασυνοριακές ή παραβάσεις. Στα πλαίσια των εμπορικών διαπραγματεύσεων φυσικά έχουμε πλήρη συνέστηση του θέματος αυτού και στο TTIP και σε άλλες διαπραγματεύσεις, Μερκοζούρ, Ιαπωνία, πάντα θα το λαμβάνουμε υπόψη. Θα κάνουμε πολλή προσπάθεια για τις γεωγραφικές ενδείξεις, τις ενδείξεις γεωγραφικής προέλευσης. Επειδή είναι πολύ σημαντικό βέβαια ο εινικός τομέα για την Ελλάδα και την Ευρώπη βέβαια. 60% της παγκόσμιας παραγωγής στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Θα είναι λοιπόν πολύ σημαντικό θέμα όπου δεν θα υποχωρήσουμε έναντι των ΗΠΑ ή ή ουδήποτε άλλου στις διαπραγματεύσεις. Οι γεωγραφικές ενδείξεις προέλευσης είναι πολύ σημαντικό μέτρο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βοτσεχόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, δέκα δευτερόλεπτα αφιερώσατε στην ομιλία σας στο θέμα του ρωσικού εμπάργου. Ενώ το πρόβλημά μας είναι τεράστιο και η κρίση βαθύτατη εξαιτία του εμπάργου που εφάρμοσε η Ρωσία. Ιδιαίτερα σε γειτονικέ χώρε τη Ρωσία, όπω είναι η Φιλανδία, οι χώρε τη Βαλτική και η Πολωνία. Ερωτώ λοιπόν, θα χρησιμοποιήσετε το αποθεματικό εκτάκτο ανάγκης με βάση το άρθρο 25 του κανονισμού 1306. Νομίζω ότι είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση αυτού του αποθεματικού κρίση εκτάκτου ανάγκη. Ε, και το συζητήσαμε αυτό και στην τελευταία ολομέλεια του Στρασβούργου. Είμαστε υπέρ αυτή τη ενεργοποίηση. Εσεί τι γνώμη έχετε. Γιατί οι Πολωνοί αγρότε δεν έχουν ε, λάβει ούτε ένα ευρώ μέχρι στιγμής ως αποζημίωση. Καταρχήν θα ήθελα να σας ε, διευκρινίσω ότι τα μέτρα ε, για τις κρίσεις ε, θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του 2015, όχι το 2014. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν το ευρύτερο δημοσιονομικό πλαίσιο και θα γνωρίσουμε μέχρι τις 15 Οκτωβρίου ποιες είναι οι τελευταίες προβλέψεις ε, δεδομένου και του ρωσικού εμπάργου και ποια θα είναι η οικονομική επιβάρηση για το 2015. Και μάλιστα στο Μιλάνο το Συμβούλιο Υπουργών συζήτησε αυτό το θέμα αλλά δεν κατέληξε συμφωνία για τις ε, συμπληρωματικές ενισχύσεις. Πάντως, ε, ο Επίτροπος Τσόλος ε, εξήγηλε 165 εκατομμύρια ευρώ συμπληρωματική ενίσχυση. Το αποθεματικό αυτό εκτάκτο ανάγκης δεν αφορά μόνο τους αγρότες, γιατί αν αφαιρέσουμε χρήματα αυτό το αποθεματικό είναι σαν να τα αφαιρούμε από τις όλων των γεωργών. Ε, το θέμα αυτό αφορά μια απόφαση γεωργικής πολιτικής. Θα συνεργαστώ λοιπόν και με τους υπόλοιπους επιτρόπους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προασπίσουμε αυτό το αποθεματικό και με βάση τις ε, αποφάσεις γεωργικής πολιτικής που ελήθηκαν και τα μέτρα ενεργοποίησης να χρηματοδοτηθούν από ειδικά κονδύλια. Bardzo, bardzo dziękuję. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ρόντε. Δεν ξέρω τι να πω κύριε Χόγκαν. Να βάλω την πρώτη μου ερώτηση που δεν απαντήσατε για την εφαρμογή ή να προχωρήσω σε μια άλλη σημαντική ε, ερώτηση. Θα κάνω το δεύτερο αλλά θα αντιμετωπίσετε την πρώτη μου ερώτηση κάθε φορά που θα συναντιόμαστε τα επόμενα πέντε χρόνια. Τώρα, το άνοιγμα των νέων αγορών, αυτή είναι η δεύτερη ερώτησή μου, είναι πάρα πολύ σημαντική. Εμείς στο Υπουργείο Γεωργίας στη Δανία και σε άλλες ε, υπηρεσίες να μην χρησιμοποιούμε τους υπαλλήλους μας μόνο σαν ελεγκτές, αλλά και σαν πρέσβης για τον γεωργικό τομέα. Και έτσι βοηθάμε τον τομέα της γεωργίας να μπαίνει και σε νέες αγορές. Αυτό ακριβώς χρειάζεται να κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην παρούσα κατάσταση. Είσαστε λοιπόν διατεθειμένος να καλλιεργήσετε ένα νέο πνεύμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου οι υπάλληλοι να παίζουν ένα δραστήριο ενεργητικό ρόλο και όχι απλά να είναι ελεγκτές και να λειτουργούν αμυντικά. Φυσικά και ναι. Φυσικά και εγώ θα πάρω ένα τέτοιο ρόλο, θα αναλάβω ένα τέτοιο ρόλο προσωπικά και το ίδιο και οι υπηρεσίες μου για να πολλαπλασιάσουμε τις αγορές μας να δούμε τι δυνατότητες έχουμε μετά από τις κρίσεις στη Μέση Ανατολή και στην περιοχή της Ουκρανίας-Ρωσίας. Όλοι ε, θα πρέπει να ε, πάρουν μέρος στην προσπάθεια αυτή. Υπάρχει φυσικά ανάγκη και για καλύτερο συντονισμό σε σχέση με την προώθηση της πρόσβασής μας στις διεθνείς αγορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κυνηγάμε με κάθε κόστος την επιτυχία αλλά σε ιδιαίτερες δύσκολες ε, πολιτικά περιοχές θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που μας δίνει η απελευθερωμένη μας αγορά. Και έχουμε και το δίκτυο ασφαλείας και τα μέσα, ε, ιδιαίτερα τα λεγόμενα μικρομέτρα, micro measures, τα οποία θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τα επιμέρους προβλήματα. Ε, τώρα για τα επόμενα χρόνια έχουμε ε, για τέτοιου είδους μέσα τουλάχιστον 30 εκατομμύρια και έτσι θα βοηθήσουμε νομίζω να ανοιχτούν και καινούργιες αγορές για τα προϊόντα μας. Ευχαριστώ. Κύριο Κάρθη. Υποψήφια Επίτροπε, ξέρουμε τι είπατε για τα άτομα που έκαναν αιτήσει για κοινωνικές κατοικίες όταν ήσασταν υπουργό στέγασης. Μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε πόσοι πολιτικοί αντίπαλοι και πόσοι δημοσιογράφοι διαφόρων μέσων ε, της αντιπολίτευσης έλαβαν ε, γράμματα από δικηγόρους από σας και γιατί επίσης αποφασίσατε να σταματήσει κάποια μελέτη που είχε ε, ξεκινήσει ο προκάτοχός σας για παρατυπίες σε σχέση με την χωροταξία. Επίσης ε, ακούθηκε, ακούστηκε ότι υπάρχουν παρατυπίες μεγάλου ύψους για κάποιες ε, ε, από τις δραστηριότητές σας. Επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο λοιπόν και μάλιστα έχουν ξεκινήσει κάποιες δικαστικές διαδικασίες εναντίον σας, πιστεύετε ότι θα έχετε το χρόνο και την δυνατότητα να αφοσιωθείτε στα καθήκοντά σας ως Επιτρόπου. Πρώτον, ξέρω ότι είστε νέος κοινοβουλευτικός, αλλά Ήμουν 27 χρόνια μέλος του Εθνικού Κοινοβουλίου. Ξέρω ότι είναι κοινοβουλευτικό προνόμιο και τι όχι. Και βεβαίως, ε, ε, αν γίνεται κάποια προσπάθεια δυσφήμισης πολιτικών, έχουν κάθε δικαίωμα να αμυνθούν. Και είπα, θα συνεργαστώ πλήρως με την Επιτροπή για διαφάνεια, ε, αναλογικότητα και οτιδήποτε έχει να κάνει με τον προπολισμό της Ένωσης. Δεν σταμάτησα καμία έρευνα άλλος υπουργός ήταν υπεύθυνο για τη διεξαγωγή της. Άρα ε, σε λάθος άτομα απευθύνεστε, λάθος στιγμή. Τα 50 εκατομμύρια ε, ευρώ του, ευρω... του... της εταιρείας Ιρλανδικό Ίδωρ ήταν αυτά που χρειαζόντουσαν για ε, την υποδομή και τη λειτουργία της και χρειαζόντουσαν για να δώσουμε καλύτερη ποιότητα ύδατος. Εάν δημιουργεί κανείς ένα νέο σύστημα πρέπει να δαπανίσει ε, τα αναγκαία ποσά. Και η ρυθμιστική αρχή για την ενέργεια θεωρεί ότι από τα 180 εκατομμύρια που δαπανήθηκαν σε αυτή την προσπάθεια, 172 δαπανήθηκαν σωστά. Ξέρω ότι είστε κατά τη Ευρώπη και είστε και κατά τη υποψηφιότητά μου. Αλλά έλαβα ένα θαυμάσιο γράμμα από τον συνάδελφό σα, τον Υπουργό Γεωργία στη Βόρεια Ιρλανδία, που είναι μέλο του Sinn Féin. Αγαπητέ Φιλ, σε συγχαίρω για την ε, πρόταση που έχει γίνει να γίνει ε, Επίτροπο Γεωργία είναι ε, υψηλού κύρου ε, αρμοδιότητα. Θα βοηθήσει και εθνικά και θα ήθελα να σα δω όταν αναλάβετε τα καθήκοντά για να συζητήσουμε τομεί αμοιβαίου συμφέροντο για να έχουμε ουσιαστική ε, σχέση συνεργασία. Ξέρω πόσο σημαντική είναι η γεωργία στο Βορρά. Το μόνο λοιπόν που μπορώ να πω είναι ότι δεν υπάρχει αρκετή πειθαρχία εντό του Σινφέιν. Ελπίζω να μην σας δημιουργήσει προβλήματα λοιπόν αυτό που είπατε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ροπέ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε υποψήφιε Επίτροπε, έχετε αναγγείλει ενδιάμεση επανεξέταση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Θα πρέπει εν ώψη αυτής ενδιάμεσης ε, επανεξέτασης να γεφυρώσετε το, το χάσμα των πληρωμών που υπάρχει μεταξύ των γεωργών στα διάφορα κράτη-μέλη. Το ανέφερε και ο πρόεδρος Γιούνκερ. Γιατί οι πληρωμές στη Ρουμανία ή στις βαλτικές χώρες είναι πολύ χαμηλότερες από το μέσο όρο πληρωμών στους γεωργούς. Ενώ το κόστος της γεωργίας στις βαλτικές χώρες ε, είναι εξίσου υψηλό και μάλιστα το ενεργειακό κόστος είναι ακόμη πιο υψηλό στις χώρες αυτές τεχνολογία είναι πιο δαπανηρή και όλα αυτά αυξάνουν το κόστος παραγωγής στην Βαλτική Γεωργία. Γι' αυτό και υστερούμε τόσο πολύ. Η μισθή μάλιστα είναι ακόμη χαμηλότερη και δημιουργείται έτσι ένας φαύλος κύκλος. Στην εισαγωγική σας ομιλία δεν μιλήσατε για την πανόλη των χείρων, ένα σοβαρότατο πρόβλημα, σοβαρότατη ε, επιζώτη που παρουσιάζει έξαρση, μάλιστα σε πολλές χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όντω, ε, η κοινή υγειορική πολιτική είναι ένα σημαντικό βήμα προ σωστή κατεύθυνση σε ό,τι αφορά την εσωτερική και εξωτερική σύγκληση και θέλουμε πιο ακριβωδίκη κατανομή των ε, γεωργικών ενισχύσεων μεταξύ των χωρών και μεταξύ των γεωργών. Και φυσικά έχει ε, μειωθεί ο σύνδεσμό με τα ιστορικά σημεία αναφορά. Θα πρέπει βέβαια να επιτύχουμε τι αρχέ προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Στόχου. Έχουν γίνει όμως ε, σημαντικές αλλαγές από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και πιστεύω ότι έχουμε κάνει πρόοδο για πιο ακριβωδίκη κατανομή των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των περιφερειών. Η αυτονομία και η ελαστικότητα που δώσαμε στα κράτη-μέλη θα βοηθήσει τους ε, μικροκαλλιεργητές, ε, τους αγρότες σε ορεινές ή απόμακρες περιοχές και θα γεφυρωθεί έτσι το χάσμα των πληρωμών. Φυσικά θέλουμε μια βιώσιμη γεωργία, ένα βιώσιμο γεωργικό κλάδο. Θέλουμε μεγιστοποίηση του βασικού τουλάχιστον εισοδήματο και αύξηση των ε, ευκαιριών για πρόσβαση στην αγορά. Το 69% των ε, γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι μικρότερες από 5 εκτάρια. εκτάρια. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα βέβαια σε πολλές περιοχές, αλλά πιστεύω ότι με τις μεταρρυθμίσεις ε, θα δούμε σε κάθε κράτος μέλος τι μηχανισμός έχει χρησιμοποιηθεί και φυσικά στην ενδιάμεση επανεξέτηση θα τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη και θα διδαχθούμε από τα λάθη μας. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μπονάνο. Ε, Κύριος Μπονάνο, συγγνώμη. Συγγνώμη, λάθος. Η κυρία Μόη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κοινή αγροτική πολιτική έτσι όπως έχει σχεδιαστεί από την Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο δεν επηρέασε θετικά Διαφθορά και οργανωμένη εγκληματικότητα έχουν ελέγξει σε πολλές χώρες τις άμεσες πληρωμές ε, όπως και στην ε, Ιταλία. Διάφορα λόμπι γεωργικά μαζί με πολιτικούς και τοπικούς συμβούλους εκμεταλλεύτηκαν τις δυνατότητες που είχαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις διάφορες περιοχές. Πώς θα λύσετε το πρόβλημα αυτό. Οι άμεσες πληρωμές πώς θα ελεγχθούν. Ποιος θα δώσει εγγυήσει ε, έτσι ώστε τα πρότυπα διανομής των πιστώσεων αυτών να μην υποκύπτουν σε συμφέροντα πελατειακά και εγκληματικά όπως σήμερα στην Ιταλία. Υπάρχει ένα δίκτυο κυρώσεων εις βάρος τέτοιου είδους καταχρήσεων πώς θα προστατεύσετε από τις απάτες της εθνικές ε, παραγωγές όπως το λεγόμενο Made in Italy. Δεν γνώριζα για τις δυσκολίες αυτού του τύπου σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων στην Ιταλία για λόγους ε, πίεσης πολιτικούς και ποινικού. Φυσικά θα ενδιαφερθώ και θα μάθω περισσότερα για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Αλλά αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει η κοινή αγροτική πολιτική είναι να βρει έναν τρόπο να διαθρέψει φυσικά πρώτα τον ευρωπαϊκό πληθυσμό και τον υπόλοιπο κόσμο. Επίσης λόγω της μεγάλης πίεσης που θα υπάρξει στο μέλλον λόγω ακριβώς της αύξησης του πληθυσμού και των περιβαλλοντικών περιορισμών γνωρίζουμε την, ε, την σπανιότητα ορισμένων πόρων και θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Και γι' αυτό βοηθάμε τα κράτη-μέλη στα πλαίσια της αρχής της επικουρικότητας να διαχειριστούν τέτοιου είδους θέματα. Φυσικά δεν υπάρχει μαγική συνταγή και η ευελιξία η οποία υπάρχει και στα πλαίσια της γεωργικής παραγωγής και στα πλαίσια των προγραμμάτων για την ανάπτυξη της υπαίθρου ε, νομίζω ότι θα βοηθήσουν και θα υπάρξει μια υπηρεσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θα συνδράμει και την Ιταλική Διοίκηση. Και φυσικά αν υπάρχουν περαιτέρω θέματα θα είμαστε στη διάθεσή σας. Και τώρα ήρθε η ώρα του κυρίου Μπονάνο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ομιλώ εκ μέρους της πιο μεγάλης οργάνωσης στον τομέα της εκτροφής ε, πτηνών και ζώων γενικότερα. Για τους νέους ε, κτηνοτρόφους ε, αλλά και τους γεωργούς, τους νέους στον τομέα των οποροκυπευτικών κτλ. Τι θα κάνετε για να τους προστατεύσετε. Τους μεγάλους τους φροντίζει η Ευρώπη, τους μικρούς τους ξεχνά και ξέρετε πόσοι νέοι γεωργοί αυτοκτόνησαν γιατί οι κανόνες που δημιουργεί η Ευρώπη δημιουργούν επιπλέον δυσκολίες οι οποίες προστίθενται στην κρίση η οποία ισοβεί στη διεθνή αγορά και στον γεωργικό τομέα. Υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες γιατί έχετε και το βάρος των προκατόχων σας με μια κοινή αγροτική πολιτική παρανοϊκή η οποία δημιούργησε τα προβλήματα του σήμερα. Εσείς ε, δεν θέλω ε, να είστε ένας παρεμβησίας Ευρωπαίος και από κάτω ουσιαστικά να είστε ασιάτης και να προωθείτε άλλα συμφέροντα. Thank you very Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως οποιαδήποτε μεταρρύθμιση θέλει χρόνο για να εφαρμοστεί η μεταρρύθμιση της κοινή γεωρικής πολιτικής. Όλοι ανησυχούν όταν υπάρχουν αλλαγές. Είναι πολιτιστικό το θέμα αυτό. Και στην Ιρλανδία έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά δεν μπορούμε να μην κινηθούμε. Η κατεύθυνση της ε, ΚΚΠ από το 92 και μετά είναι απομάκρυνση από την στήριξη της, ε, των τιμών προς, την προς τη στήριξη του εισοδήματο. Πρέπει λοιπόν να το κάνουμε αυτό και το λαμβάνουμε υπόψη όταν έχουμε διμερείς και πολυμερείς διαπραγματεύσεις. Πρέπει να καταλάβουν όλοι πόσο μπορεί να συμβάλλει η Ευρώπη στην επιστημιστική ασφάλεια στο μέλλον. Διατηρώντας λοιπόν βιώσιμες εκμεταλλεύσεις με τη βασική ενίσχυση εισοδήματο που δίδεται από τη μεταρρύθμιση διατηρώντας ε, την, διατηρώντας την ε, περιβαλλοντική επίσης ε, διάσταση και με την ενίσχυση που δίνουμε μέσω διαφόρων μέτρων στην αγορά θα διασφαλίσουμε ότι η Ένωση είναι ανταγωνιστική, ότι μπορεί να έχει επιτυχείς εμπορικές σχέσεις και να ανοίξει και νέες αγορές σε άλλες περιοχές από αυτές που είχαμε τώρα και που είναι σε κατάσταση σειράξεων όπως ε, η Ουκρανία, η Ρωσία και η Μέση Ανατολή. Να δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει η μεταρρύθμιση στην πράξη και μετά σε ένα-δύο χρόνια θα δούμε τι περαιτέρω αλλαγές ενδεχομένω χρειάζονται για περαιτέρω βελτίωση. Ευχαριστώ. Περνάμε στον τρίτο γύρο. Πρώτος ομιλητής του τρίτου γύρου, ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ αγαπητέ υποψήφιε το αποτέλεσμα της τελευταίας μεταρρύθμισης για μένα είναι έτσι και έτσι. Ε, λίγα χρήματα παραπάνω αλλά περισσότερη γραφειοκρατία. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω τι συγκεκριμένα βήματα σκοπεύετε να λάβετε για να μειώσετε την γραφειοκρατία και να πλουστεύσετε την ΚΓΠ. Ε, πώς θα γίνει το πρασίνισμα στον πρώτο πυλώνα στην ε, επανεκτίμηση πρέπει να το συζητήσουμε. Και τις προτάσεις του αγαπητού συναδέλφου, τις πέντε προτάσεις του συναδέλφου Άλμπερντες θα τις κοιτάξετε, ήταν σε ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Γιατί θεωρώ ότι τις προτάσεις μας ε, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεν τις έλαβαν επαρκώς υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, Υπάρχει η αντίληψη ότι πρέπει να επιδιώξουμε καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών και του Κοινοβουλίου. Και συμφωνώ απόλυτα το θέμα αυτό και θέλω να είμαι σε επαφή με την ηγεσία των ομάδων για να βελτιώσουμε την επικοινωνία. Εγώ 32 χρόνια είμαι εκλεγμένος, καταλαβαίνω λοιπόν τους ε, πολιτικούς, καταλαβαίνω ότι πρέπει να ενημερώνετε του ψηφοφόρου σα για την εφαρμογή των μέτρων αυτών με πολύ διαφανή και ειλικρινή τρόπο. Υπάρχουν διοικητικοί κανόνε που ρυθμίζουν ε, την ε, σχέση μεταξύ του ιδιαίτερου γραφείου μου και των υπηρεσιών. Η νέα Επιτροπή γενικά θα έχει νέου κανόνε, Θα πρέπει να δούμε πώ θα συνεργαστούμε. Παρατήρησα ότι στους ειδικού ε, τομείς πολιτικής υπάρχει περιθώριο συνεργασίας με την Επιτροπή Γεωργίας θα έπρεπε να μπορεί να συμμετάσχει περισσότερο στην φάση διαμόρφωσης προτάσεων. Δεσμεύτηκα ότι στην αρχή της θητείας μου ήδη, πολύ στην αρχή, θα κάνουμε μία εξέταση screening της ΚΚΠ για να την απλοποιήσουμε. Αλλά όπως είπα η απλοποίηση δεν είναι απλή υπόθεση. Θα προσπαθήσουμε με βάση και τα παραδείγματα που θα μου δώσετε από τη χώρα σας να επιδιώξουμε το πρασίνισμα. Τον περασμένο Απρίλιο δηλώσαμε ότι θα εξετάσουμε το πρασίνισμα, να δούμε τις περιοχές οικολογικής εστίασης. Όταν θα έχουμε επαρκή στοιχεία, θέλουμε να κάνουμε μια πολύ εμπεριστατωμένη αποτίμηση της κατάστασης να λάβω υπόψη και την εκθεσιντές, όλες τις προτάσεις που έχουν γίνει, όλα όσα μου έχετε ήδη πει για την συγκεκριμένη εφαρμογή στο επίπεδο κάθε κράτους μέλους. Τα κράτη-μέλη όμως πρέπει να συνεργαστούν με την Κομισιόν ούτως ή άλλως με την Επιτροπή για την Εφαρμογή της ΚΑΠΑΓΑΜΑΠΗ και θα δώσω τα μέσα στην Επιτροπή για να το κάνει. Σας ευχαριστώ. Η ε, κυρία Αγγιλέρα. Κύριε Χόγκαν. Οι εμπορικές πρακτικές, οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές ε, δημιουργούν συστημική ανισορροπία στην αλυσίδα τροφίμων. Τα συστήματα ε, συμβάσεων που προτείνει η ενιαία ΚΟΑ δεν, δεν αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τι πρωτοβουλίες θα αναλάβετε απέναντι στις, ε, στους συναδέλφους του ανταγωνισμού για να βελτιώσετε τη θέση των γεωργών στην επιστηστική αλυσίδα. Δύο είναι οι βασικοί τόμοι ε, για την ε, Γεωργία του Νότου. Ελαιόλαδο και οπωροκυπευτικά. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τον κοινωνικό ιστό των ε, περιοχών παραγωγών. Τα απορροκυπευτικά λειτουργούν καλά, δεν απαιτούν μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Πώς θα βελτιώσετε την ανταγωνιστικότητα όμως στον τομέα αυτό που μερικές φορές χρησιμοποιείται στις εμπορικές συμφωνίες ως αντιστάθμισμα και τι θα, γίνεται, τι θα γίνει με το ελαιόλαδο, θα, θα συνεχίσετε το σχέδιο δράσης για το ευρωπαϊκό ελαιόλαδο που ξεκίνησε ο προκάτοχός σας πριν από μια διετία. Σας ευχαριστώ. Συμμερίζομαι πλήρως ε, τα σχόλια της συναδέλφου Μάλμστρομ ότι οι εμπορικές ε, πρακτικές και συμφωνίες θα αποτελέσουν ε, σημαντική συνεισφορά στην ανάκαμψή μας. Γι' αυτό χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια και συμφωνώ με την έκκλησή της για αποκατάσταση της διαφάνειας. Και μάλιστα θα δημοσιεύσουμε και καταλόγους ε, ε, και θα δημοσιεύσουμε όλες τις σχετικές ε, συμφωνίες διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του TTIP και ελπίζω και οι Ηνωμένε Πολιτείε να κάνουν το ίδιο για να μην έχουμε καμία εμπιστευτικότητα να, απο... να αποκατασταθεί η διαφάνεια και να ξέρουν όλοι τι διαμείβεται στις διαπραγματεύσεις του TTIP. Φυσικά υπάρχει μεταρρύθμιση και προ... προτείνονται άμεσα ενισχύσεις ε, και στα πλαίσια της αγροτικής ε, ανάπτυξης ε, και μεγαλύτερη υποστήριξη στους οργανώσεις παραγωγών. Και σίγουρα η νέα μεταρρύθμιση θα προσφέρει καλύτερη ολοκλήρωση των ενισχύσεων, ιδιαίτερα στα οποροκυπευτικά. Για το ελαιόλαδο δεν είναι ο τομέας που γνωρίζω καλύτερα, αλλά εξοικειώνομαι όλο και περισσότερο. Και κυρία Γκαρσία, ε, προσβλέπω στη δική σας ενημέρωση και διαφωτισμό στις επαφές που θα έχω με τους διαφερόμενους του κλάδου για να ενημερωθώ καλύτερα για τα προβλήματα των ε, ελαιοπαραγωγών στο Νότο. Η κυρία Κοσεύσκα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Χόγκαν, επειδή έχω ε, συν πολύ λίγο χρονικό διάστημα, θα ήθελα να επικεντρωθώ σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πιστεύετε ότι υπάρχει δυνατότητα αύξηση των άμεσων ενισχύσεων για τους Πολωνούς για την ε, επόμενη περίοδο προγραμματισμού μέχρι το 2020 και λαμβάνοντας υπόψη τις ε, ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες και τι γίνεται με το ρωσικό εμπάργο και την κρίση που δημιουργήθηκε στα τρόφιμα θα αντιδράσετε άμεσα και αποτελεσματικά προκειμένου να αντισταθμίσουμε τις τεράστιες απώλειες των γεωργών. Επίσης, για τις ε, γαλακτοκομικές ποσοστώσεις, είστε υπέρ της αποκατάστασης της επιστροφής ε, των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων και τι θα γίνει με την τελευταία αυτή φάση. Σε ό,τι αφορά την επιζωτία το, της των χείρων, κυρίως από την Αφρική, γιατί είχαμε τεράστιες ε, αποζημιω... τεράστιες απώλειες για τους γεωργούς από το θέμα της πανόλης των χείρων και τι... ποια είναι η γνώμη σας για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα. Δύσκολο να δώσω απαντήσεις σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. δεν θα λύσω όλα τα προβλήματα στα οποία αναφερθήκατε τα επόμενα πέντε χρόνια, αλλά η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ θα βοηθήσει πολύ σε επίπεδο ε, σύγκλησης. Ας μην ξεκινήσουμε ξανά την τελευταία συζήτηση η οποία οδήγησε στη μεταρρύθμιση τα προηγούμενα χρόνια. Πάντως στα πλαίσια της ενδιάμεσης αναθεώρησης θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να διατηρήσουμε ε, βιώσιμες μεσαίες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ξέρετε ότι ένα μεγάλο ποσοστό είναι μέχρι 15 εκτάρια 5 συγγνώμη, εκτάρια και ταυτόχρονα με τα προγράμματα στήριξης των εισοδημάτων θα μπορέσουν τα κράτη-μέλη να αυτονομηθούν εν πολλής και η δική σας χώρα έχει αυτή τη δυνατότητα για να μπορέσει να στρέψει κάποιους πόρους σε συγκεκριμένους τομείς οι οποίοι συγκυριακά στις διάφορες περιοχές υφίστανται έκτακτες πιέσεις. Ε, έχετε στραφεί σαν Πολωνία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχετε δει τι μέσα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν οι ανάγκες των γεωργών για τους οποίους ανησυχείτε. Ε, και η στήριξη μέσω άμεσων πληρωμών θα βελτιωθεί σε σχέση με το παρόν καθεστώς και θα είμαστε το 2020 σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι σήμερα. Είμαι υπέρ της κατάργησης των ποσοστώσεων στα γαλακτοκομικά. Τα μέσα της αγοράς είναι εκεί για να διασφαλίσουν τη σταθερότητα της αγοράς και να λύσουν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια όπως το εμπάργο προς τη Ρωσία. Συνειδητοποιώ τις τεράστιες δυσκολίες τις οποίες αντιμετώπισαν οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ε, λόγω ακριβώς του εμπάργο προς τη Ρωσία και ο Επίτροπος Σιόλος μέσω στοχευμένη στήριξης προσπάθησε για να βρει λύσεις. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος um, Ευχαριστώ κύριε υποψήφιε επίτροπε. Η πει να πρέπει να στοχεύσει περισσότερο στην ε, καινοτομία και να βοηθήσει την επιχειρηματικότητα. Αν δεν το κάνουμε αυτό θα χάσουμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Οι καινοτόμοι γεωργοί αντιμετωπίζουν προβλήματα συχνά γραφειοκρατίας. Για παράδειγμα αυτή η οδηγία για τα νετρικά. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπάρχει όριο για τα νετρικά αλλά τα στα ε, υπόγεια ύδατα, αλλά θα πρέπει να είναι ευθύνη του Γεωργού πώς θα συμμορφωθεί. Γι' αυτό δεν είναι δυνατόν να μην ε, έχουν δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν πάνω από 170 κιλά ε, φυσικής ε, κοπριάς ανεκτάριο. Δεν μπορεί ένας γεωργός να χρησιμοποιήσει την κοπριά του, αλλά επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τεχνητά λοιπάσματα αντί γι' αυτό. Παρακαλώ, μπορείτε να μας δώσετε τρία παραδείγματα πώς θα μειώσετε τη γραφειοκρατία για να βοηθήσουμε την επιχειρηματικότητα. Και δεύτερον, τι θα κάνει ο υποψήφιος επίτροπος, ούτω ώστε να ε, λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον των γεωργών εντός του κολεγίου των επιτρόπων. Η χρηματοδότηση της ΚΑΜΑΓΑΜΑΠΗ και της γεωργίας έχει μειωθεί, όπως υπόθηκε, αλλά είναι ακόμη πολύ σημαντικό τμήμα του ενωσιακού προπολογισμού, 38% του συνολικού προπολογισμού. Είναι λοιπόν ένα πολύ μεγάλο τμήμα για να δημιουργηθούν ε, θέσει εργασίας, ε, ανάπτυξη της υπαίθρου, επισητιστική ασφάλεια. Και ο κεντρικός ρόλος ε, των τροφίμων δεν αμφισβητείται. Είδαμε τι προβλήματα έχουν οι κατασκευές και άλλοι τομεί όπου οι κάτοικοι της υπαίθρου μπορούσαν να βρουν δουλειά. Τώρα λοιπόν εξαρτώμεθα όλο και περισσότερο από την ε, επιχειρηματικότητα των νέων γεωργών που επιστρέφουν σε, ε, στην Ήπεθρο και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να διαφοροποιήσουμε τις μορφές απασχόλησης. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε στους τομείς άλλων επιτρόπων για να τους βοηθήσουμε. Ορίζον 2020, επιχειρηματική βοήθεια για να βοηθήσουμε την ανάπτυξη της τα μέτρα έξω από την ε, ε, είσοδο των εκμεταλλεύσεων, όλα αυτά σημαίνουν ότι ε, δεν αξιοποιούμε μόνο το 38% αλλά και άλλα τμήματα του προπολογισμού. Ίσως έχετε κάποιες ιδέες να μας βοηθήσετε. Τώρα για την οδηγία για τα νητρικά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να υπάρξει ισορροπία μεταξύ της παραγωγικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος, της διαχείρισης και της βιωσιμότητας. 45% των ε, ε, υδατίνων πόρων μας υφίστανται πιέσεις. Φυσικά θέλουμε να βοηθήσουμε λοιπόν τα μέτρα άρδευσης, αλλά δεν κάνουμε αρκετά για να προστατεύσουμε τις πηγές ύδατος. Πρέπει λοιπόν να επιδιώξουμε μια ισορροπία. Και δεν νομίζω ότι ο Γεωργός για τα θέματα της ε, πολυτομιακής συμμόρφωσης είναι ο καλύτερος για να διασφαλίσει την πολυτομιακή πολλαπλή ε, συμμόρφωση. Πρέπει λοιπόν να εφαρμοστούν τα μέτρα που προβλέπει η οδηγία για τα νητρικά. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Φλάναγκαν. Ε, ε, welcome, Phil. Να καλωσορίσω τον Φιλ. Άκουσα ότι θέλετε να συνεργαστείτε με όλους τους πολιτικούς. Καλό είναι αυτό γιατί είχατε πει στα Ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης ότι διάφοροι σαν και εμένα και τον Κάρτη είμαστε στο περιθώριο και δεν έχουμε καμία σημασία. Αναφερθήκατε στη σύγκληση. Ε, τα κράτη-μέλη υποτίθεται θα προχωρούσαν σε ενιαίες μορφές πληρωμών ανά εκτάριο από το 18 και μετά. Ένα πρότυπο δηλαδή σύγκλησης. Αυτό σημαίνει ότι το 20% των πλουσίων, των πιο πλουσίων, θα παίρνουν άνω το 80% των ε, πληρωμών. Σήμερα ο Ιρλανδικός τρύπος λέει ότι στην ουσία προσπαθήσατε να εκφοβήσετε ε, με τους ε, υποστηρικτές σας αυτούς οι οποίοι έχουν διαφορετική άποψη. Θα ενισχύσετε τους εκατομμυριούχους και αυτούς που έχουν μεγάλες εκτάσεις ή θα κάνετε αυτό το οποίο καλείται να κάνει η ΚΑΠ. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια λέει ο κύριος Όγκαν. Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι εγώ προσπάθησα σαν αντιπρόσωπος αυτών που με εκλέγουν να δημιουργώ συνθήκες που με τη σειρά τους θα δίνουν δουλειά στον κόσμο και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά θα ήθελα να έλεγα ότι κάποιοι γνωστοί μου που έστειλαν το curriculum vitae τους στο Irish Water δεν κατάφεραν να βρουν θέση απασχόλησης. Φαίνεται ότι χάνω την επιρροή μου. Έχω λοιπόν την δυνατότητα επικοινωνίας και δεν νομίζω ότι οι μικροί γεωργοί εξαιρούνται από τις διαδικασίες. Υπάρχει σύγκληση και εσωτερική και εξωτερική. Αυτό έχει σαν στόχο η μεταρρύθμιση. Έχουμε τη στήριξη των εισοδημάτων για τους μικρούς γεωργούς θα μπορούν να παίρνουν 5.000 ευρώ επιπλέον κατ' έτος λόγω ακριβώς των σωστών ε, γεωργικών ε, πρακτικών. Και οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν προωθηθεί θα επιτρέψουν στα κράτη-μέλη ε, να δίδουν και διαφορετικού τύπου βοήθεια, επιδοτήσεις και για προϊόντα τα οποία πολλές φορές αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα συγκυριακά στις αγορές. Έχουμε την δυνατότητα και μέσω άλλων τρόπων να ενισχύσουμε τον κόσμο στη Σνήπεθρο και θα στηρίξετε ελπίζω τα μέτρα τα οποία θα προτείνουμε για να υπάρξει συνέχιση της σύγκλησης ε, στα πλαίσια των εισοδημάτων από την ΚΑΠ τα επόμενα χρόνια. Αυτός θα είναι ο στόχος μου τα επόμενα πέντε χρόνια. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σεμπαστιά έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Χόγκαν. Ζητήσατε κάποια στοιχεία, θα σας τα δώσω. Οι συμβατικοί γεωργοί υπέστησαν αύξηση 40% του τελικού προϊόντος από το 2000 μέχρι το 2010 με βάση τα στοιχεία της Γεροστάτ. Τα λιπάσματα αυξήθηκαν κατά 80%, οι ζωοτροφές κατά 30% και τα φυτοφάρμακα κατά 13%. Ποιοι καρπώνονται τα, τα κέρδη από τις αυξήσεις αυτές, σίγουρα όχι οι γεωργοί. Έχουμε νέες γεωπονικές ε, τεχνολογίες και τεχνικές ε, που θα μπορούσαν να τα κάνουν όλα αυτά δωρεάν και να συμβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος και παρόλα αυτά τα αξιοποιούμε. Θα υποστηρίξετε λοιπόν μια βιώσιμη γεωργία ή θα γίνεται ο Επίτρεπος της αγροεπιστηστικής βιομηχανίας. Μιλήσατε για τα απορριπευτικά του Νότου. Δυστυχώ είναι, πολύ απογοητευμένοι και αισθάνονται καταλελειμμένοι οι γεωργοί μας από την ΚΑΠ. Και μάλιστα τα τελευταία δεκαετία συνεχίζεται η πορεία των τιμών των απορριπευτικών προϊόντων. Εγώ είμαι πέρα τη γεωργική πολιτική, τη κοινή πολιτική. Τι θα κάνει η Ευρώπη όμω για να βοηθήσει του γεωργού για να μην μείνουν εγκαταλελειμμένοι στο έλεος του. Ευχαριστώ. Σίγουρα θα στηρίξω ένα βιώσιμο γεωργικό μοντέλο. Ήμουν ανέκαθεν υπέρμαχος αυτής της προσέγγισης και το δήλωσα και στην αρχική μου παρουσίαση και δεν μπορούμε να έχουμε μια ενεργό γεωργία χωρίς ε, καλή ποιότητα εδάφους, καλή ποιότητα ε, ύδατος και φυσικά η μεταφορά ε, της τεχνολογικής γνώσης είναι σημαντική και θα πρέπει να στηρίξουμε ταυτόχρονα την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα. Και αυτές είναι προτεραιότητες ε, και του Επιτρόπου Τσόλος. Θέλουμε να προωθήσουμε την καινοτομία στην τεχνολογία για να εξασφαλίσουμε μια βιώσιμη γεωργία. Επίσης, ε, Έχουμε συζήτηση για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι και τα μακροπρόθεσμα μέτρα, γιατί οι αηφορία της γεωργίας πρέπει να εξασφαλίσουμε. Φυσικά πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε άμεσα για να αντισταθμίσει τις απώλειες από το ρωσικό εμπάργο. Για να μην μιλήσουμε για την νομοθετική διαδικασία. Ε, προσπαθήσαμε να επιταχύνουμε την λήψη μέτρων για να ελαφρύνουμε τους γεωργούς. Ιδιωτική αποθήκευση, ε, παρέμβαση και μάλιστα τα απορροκυπευτικά βρέθηκαν στο επίκεντρο της ε, προσοχής μας, γιατί τα προκυπευτικά είναι αναλώσιμα αγαθά και ήταν αυτά που κατεξοχήν εξάγονταν προς τη Ρωσία. Οπότε λαμβάνουμε υπόψη τις ε, ιδιαιτερότητες του κλάδου και στις προτάσεις μας για το 2015 θα καλύψουμε και αυτό το τομέα και περιμένω φυσικά τις προτάσεις σας ε, και φυσικά θέλουμε πιο ολοκληρωμένη στήριξη των οργανώσεων παραγωγών. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να δεχτώ την δήλωσή σας ότι δεν έχει γίνει τίποτα για τον τομέα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Τσούλο. Έχετε το λόγο. Το κίνημα από το οποίο προέρχομαι πιστεύει ότι η Ευρώπη πρέπει να υπηρετεί τους πολίτες. Έχουμε ανάγκη από μια ομοιογενή και λειτουργική εσωτερική αγορά. Εσείς μιλήσατε για τη Γεωργία, αλλά η κρίση με την Ρωσία και αυτά τα οποία συζητάτε στα πλαίσια του TIP με τη ΣΥΠΑ δείχνουν ότι ακολουθείτε τον αντίθετο δρόμο και υπάρχει επίσης και τρομερός ανταγωνισμός ανάμεσα σε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα κάποια προϊόντα, κάτι το οποίο δεν βοηθά τη ζήτηση από πλευράς των καταναλωτών. Θα πρέπει να προστατεύουμε τους γεωργούς αλλά θα πρέπει να προστατεύουμε και τους καταναλωτές και το θέμα όταν υπάρχουν στρεβλώσεις να διορθώνονται εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων και να μην τίθεται σε κίνδυνο η παραγωγή από εξωτερικούς παράγοντες. Με λίγα λόγια, πού πάμε. Well, presently there is... Uh, Προς το παρόν υπάρχει μια ισορροπία εισαγωγών και εξαγωγών σε σχέση με τα τρόφιμα. Δεν ήταν πάντα έτσι τα πράγματα και δεν μπορούμε να προβλέψουμε απολύτως το τι θα συμβεί στο μέλλον, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, ήταν κάποτε η μεγαλύτερη εξαγωγός, μετά αμφισβητήθηκε από τη ΣΥΠΑ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το θέμα είναι το πώς θα διαποροποιήσουμε ε, την παρουσία μας σε κάποιες δύσκολες περιοχές έτσι ώστε να διατηρήσουμε το επίπεδο εξαγωγών το οποίο έχουμε μέχρι σήμερα. Η διασφάλιση προμήθειας τροφίμων είναι σημαντική όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για το σύνολο του παγκόσμιου πληθυσμού. Γιατί εμείς εν πολύ στρέφουμε ένα μεγάλο κομμάτι του παγκόσμιου πληθυσμού. Πώς λοιπόν θα ξεφύγουμε από τις προβληματικά γεωπολιτικές περιοχές ε, από τις γεωπολιτικές περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα έτσι ώστε να βρούμε λύσεις συνολικά. Ε, θα συνεργαστώ με την Επίτροπο Μάστρον πολύ στενά ε, για να συμβεί κάτι τέτοιο. Οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου του 2015 έχουν σαν στόχο να έχουμε ένα βιώσιμο σύστημα παραγωγής, βιώσιμες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, αηφορία και μέσα παραγωγής τα οποία ε, θα διασφαλίσουν τις νέες τεχνολογίες που θα μας επιτρέψουν στο μέλλον να αναπτύξουμε τα μεγέθη της παραγωγής με διαφοροποιημένο τρόπο για να καλύψουμε τις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς και μέσω συμφωνιών με τις υπόλοιπες περιοχές του κόσμου να προσφέρουμε τα κατάλληλα προϊόντα που θα έχουν ανάγκη. Ε, έχουμε επίσης και το δίκτυο ασφαλείας στην περίπτωση που υπάρχουν κρίσεις και θα υπάρχουν από καιρούς καιρών έτσι ώστε να έχουμε προστασία που χρειάζεται για τους παραγωγούς. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κέστιγκερ είπε ότι θα πρέπει να φύγει σε λίγο, γι' αυτό θα τη δώσουμε τώρα το λόγο για να προλάβει να θέσει την ερώτηση. Κυρία Κέστιγκερ. Ευχαριστώ. Είμαι συγγήτρια για τις νέες ευρωπαϊκές στρατηγικές για την ανανεώσιμα. Ξέρετε ότι η δασοκομεία είναι πολύ σημαντική για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ε, η δασοκομεία, η βιώσιμη βοηθάει και για την ανάπτυξη της γεωργίας και για την προστασία του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα τα 20 ε, εκατομμύρια ιδιωτικών ιδιοκτητών δασών παίζουν μεγάλο ρόλο. Η νέα στρατηγική για τα δάση δεν πρέπει να είναι μόνο αφηρημένη, πρέπει να βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα της δασοκομείας, να βοηθήσει την κατάρτιση και να αυξήσει την γνώση μας για την ε, πολύπλευρη σημασία του δάσους. Γι' αυτό η ερώτησή μου. Ποια κέντρα βάρους θα έχετε στο πρόγραμμα εργασίας σας για να βοηθήσετε την δασοκομεία, να βοηθήσει τη γεωργία και, το περιβάλλον. Και μπορεί η Ευρωπαϊκή Δασοκομεία να είναι σίγουρη ότι η περιφερειακή διάσταση θα γίνει σεβαστή στα πλαίσια της επικουρικότητας. Είναι πολύ σημαντικά τα δάση. Καλύπτει 50% των εδαφών μας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικός τομέας. Πολλά μπορούμε να κάνουμε. Πολλά περισσότερα για θέσεις εργασίας, για αγροπεριβαλλοντικά μέτρα που θα βοηθήσουν και τον τουρισμό σε πολλά κράτη-μέλη. Φυσικά δεν έχουμε κοινή δασική πολιτική, αλλά έχουμε στρατηγική για τα δάση χάρη στην εργασία σας ως συγκήτριας και την εργασία τη Επιτροπή. Η εφαρμογή αυτή τη στρατηγική για τα δάση θα πρέπει να είναι κοινή προσπάθεια και τη Επιτροπή και των κρατών μελών και ελπίζω ότι μπορούμε να έχουμε ένα πολιετέ σχέδιο εφαρμογή με βάση τις προτεραιότητες όπου είναι δυνατή και χρήσιμη η κοινή ενωσιακή δράση σεβόμενη την επικουρικότητα. Ο κανονισμό για τα δάση είναι το κύριο μέσο που έχουμε για να εφαρμόσουμε τη στρατηγική. Ήδη δίνει ένα συνεκτικό πλαίσιο και αρκετά μέτρα που μπορούν να μας βοηθήσουν να έχουμε βιώσιμη στήριξη των δασών ως Επίτροπος. Θα διασφαλίσω ότι ε, η ανάπτυξη των δασών παίζει τον το ρόλο της στα πλαίσια του προγράμματος ανάπτυξης υπαίθρου. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Νταντσίλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, η κοινή γεωργική πολιτική έχει λάβει υπόψη και τους νέους γεωργούς, αλλά όχι αρκετά. Η Ρουμανία, η πατρίδα μου, φαίνεται ε, στα νούμερα ότι το ποσοστό των νέων κάτω των 35 ετών που απασχολείται στη γεωργία είναι πολύ χαμηλό, μόνο 7,3%. Πώς θα ενθαρρύνετε λοιπόν τους νέους ε, να ασχοληθούν με τη γεωργία. Τι μέτρα θα θεσπίσετε για να προσελκύσουμε τους νέους στη Γεωργία και ε, να τους κρατήσουμε στην Ήπεθρο. Γιατί υπάρχει ε, αυτή η αστιφιλία που θα πρέπει να ανατραπεί. Να έχουμε ε, μετακόμιση από τα αστικά κέντρα στην Ήπεθρο. Και τι θα γίνει με τους νέους Γεωργούς. Σίγουρα ε, φροντίζεται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να να προωθήσει με 25% του συνόλου του προπολογισμού της γεωργίας στους νέους γεωργούς. Και μάλιστα θέλουμε να είναι δεσμευτικό αυτό το μέτρο με τα κράτη-μέλη και χαίρομαι γιατί τα μέτρα για τους νέους γεωργούς ε, θα βοηθήσουν άμεσα και την ύπεθρο να επιβιώσει. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό το θέμα γιατί η γεωργία έχει ε, δίνει πολλές ευκαιρίες και δυναμικό. Περισσότερο από το στεγαστικό τομέα ίσως. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους νέους να ε, αναλάβουν ηγετικό ρόλο στη γεωργία. Και θα πρέπει να τους προσελκύσουμε γι' αυτό και καλό θα ήταν ε, να ενισχύσουμε και τις γεωπονικές σχολές ώστε να προσελκύσουμε τους νέους στη γεωργία. Και αν λάβουν 25% επιπλέον για την πρώτη πενταετία οι νέοι γεωργοί, που είναι υποχρεωτικό πια, ε, πιστεύω ότι θα έχουν περισσότερα κίνητρα για να ασχοληθούν με τη γεωργία. Και μάλιστα στο νέο πρόγραμμα ανάπτυξη πέθρου έχουμε επίσης ε, για πρώτη φορά μέτρα για τη στήριξη των νέων γεωργών. Και αυτό το πρόγραμμα δίνει ευκαιρία λοιπόν για τους νέους γεωργούς. Οπότε, αν πολύ περισσότεροι νέοι έχουν πρόσβαση σε χρηματοοικονομική υποστήριξη και μπορούν να συγχρηματοδοτήσουν ε, κάποια προγράμματα και χάρη στο, στην οδηγία για την αγροτική ανάπτυξη, ε, πιστεύω ότι πολλοί νέοι θα στραφούν στη Γεωργία και με την ε, ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και με τα κοινοτικά θεσμικά όργανα προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε κονδύλια για να βοηθήσουμε νέους ε, και να τους προσελκύσουμε στη γεωργία υπέρ της κοινωνικής συνοχής και υπέρ της επιβίωσης της υπαίθρου και των αγροτικών περιοχών. Σας ευχαριστώ. Η κυρία... Ο κύριος Νίκορσον, ο συντονιστής μας, αντικαθιστά την κυρία Γκέρλινγκ. Πολύ συγκεκριμένη ερώτηση για το CPID. Είναι πολύ σημαντικό για τους γεωργούς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης ε, είναι και μία ανησυχία που έχουμε για, την, ε, ε, για τις κυρώσεις που επιβάλλονται όταν χάνουν τις ετικέτες. Κατά πόσον είναι δηλαδή αναλογικές αυτές οι κυρώσεις. Μπορείτε παρακαλώ να προσέξετε το θέμα αυτό, να ακούσετε τους γεωργούς και όχι μόνο τους υπαλλήλους σας και να βρείτε μια λύση, μια για πάντα, στην μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση. Θα συνεργαστώ με εσά κύριε Νίκολσον και με άλλου που έχουν αυτό το πρόβλημα. Είναι φαίνεται ιδιαίτερα για το Ηνωμένο Βασίλειο πρόβλημα. Ιδιαίτερα το ότι χάνονται οι ετικέτε των προβάτων. Η DG Senko, η Γενική Διεύθυνση Senko, έχει μεγάλο ρόλο όσον αφορά την μετακίνηση των ε, εκτρεφωμένων ζώων, ιδιαίτερα σε περιοχέ που τι ξέρουμε, ε, μεταξύ της Δημοκρατίας και της Βορείου Ιρλανδίας επειδή ακριβώς είχαμε προβλήματα με τα πρόβατα που χάναμε όταν μετακινούνταν. Είχαμε τέτοια προβλήματα από το 1996. Πολλά έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, ίχνη λασιμότητα, για τις ε, προδιαγραφές. Κανείς πιστεύω δεν θεωρεί ότι πρέπει να μειωθούν οι προδιαγραφές γιατί μας δίνουν και ευκαιρίες διάθεση στην αγορά και καλύτερα ανταγωνιστικότητα και καλύτερα τρόφιμα για τους καταναλωτές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους παραγωγούς. Αυτές οι ετικέτες στα ζώα φυσικά πρέπει να συζητηθούν στα πλαίσια της μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μίλλερ. Η Ευρωπαϊκή Γεωργία και η Δασοκομεία είναι σημαντικός παράγον για την απασχόληση και το εισόδημα στην Ήπεθρο. Πολλές θέσεις εργασίας τους ε, επιπλέον ε, τομείς που είναι πριν και μετά διατηρούνται επίσης. Αλλά υπάρχει τρομεγρή αφιοκρατία. όλο και περισσότερα καθήκοντα. Οπότε μικρές οικογενειακές ε, εκμεταλλεύσεις έχουν υπερβολικές απαιτήσεις και πολλές φορές τα παρατάνε. Θα απλοποιήσετε λοιπόν τις διοικητικές διαδικασίες. Θα λάβετε υπόψη τα συμφέροντα των επιχειρήσεων αυτών μέσω στόχων που υπάρχουν στα διατομιακά προγράμματα όπως το Natura 2000 ή στην οδηγία για τα νετρικά θα υπερασπιστείτε τα συμφέροντα των γεωργών έναντι άλλων γενικών διευθύνσεων και επιτρόπων. Τι θα κάνετε, ούτω ώστε η μελλοντική γεωργική πολιτική να θέσει σε πρώτη θέση την παραγωγή τροφίμων και να διατηρηθεί η γεωργική ιδιοκτησία. Βέβαια, αν θέλουμε να προωθήσουμε την επισητιστική ασφάλεια, θα πρέπει να δώσουμε ενάψματα στους παραγωγούς και ταυτόχρονα να προσφέρουμε ευκαιρίες για διαφοροποιημένες αγορές, ιδιαίτερα στους ευαίσθητους τομείς. Και, όπως είπα και προηγουμένως, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι η μόνη λύση. Γιατί αν έχουμε προβλήματα στο έδαφος και αν έχουμε προβλήματα στους υδροφόρους ορίζοντες, δεν μπορούμε να προσβλέπουμε σε αύξηση της παραγωγικότητας και σε ασφάλεια των τροφίμων. Θα πρέπει να βρούμε μία ε, ισορροπία στην πράξη. Εγώ είμαι πρακτικός άνθρωπος και θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Βέβαια μερικοί τομείς προοδεύουν πιο γρήγορα από άλλους, αλλά βασική μου προτεραιότητα είναι η απλούστευση. Θα πρέπει να μειώσουμε την γραφειοκρατία, να πλουστεύσουμε την νομοθεσία και τους κανονισμούς στο ρυθμιστικό πλαίσιο, χωρίς όμως να διακυβεύουμε τις πολιτικές και τη χρηστή οικονομική διαχείριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι με όλα αυτά θα καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις. 40% του προϋπολογισμού της, περιφερειακής, της, της αγροτικής ανάπτυξης αφιερώνεται σε περιβαλλοντικά μέτρα και ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η πορεία και να αυξηθεί. Σας ευχαριστώ. Το, ρόλο, το λόγο έχει τώρα ο κύριος Γλέζος. Πρώτη ερώτηση. Στην Ελλάδα με τη χλωρίδα των 6.000 και πλέον ειδών τα χίλια είναι ενδυμικά όπως π.χ. η μαστίχα της Χίου, η σταφίδα της Κορίνθου, το σταμναγκάθι και το δίκταμο της Κρήτης. Στην Άξο εκτός από τις πατάτες ευδοκιμή και το κίτρο. Κατ' εντολή όμως της Μέρκελ μας έφεραν ένα ψεύτικο φυτό με σιδερένιες ρίζες και γυάλινα άνθη, τα φωτοβολταϊκά. Γέμισε η Ελλάδα με αυτό το σιδερένιο φυτό που εκτόπισε καλλιέργειες που μας εξασφάλιζαν ελαιόλαδο, οποροκευτικά και σιτηρά τι θα κάνετε για να επανέλθει η καλλιεργήσιμη γη στον προορισμό της, θα έρθείτε μαζί να ξεριζώσουμε αυτό το σιδερένιο φυτό. Δεύτερη ερώτηση. Ως υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ιρλανδία κάνατε μεταρρυθμίσεις που οδήγησαν στη μείωση των κονδυλίων για το πρόγραμμα Leaders. Τι θα κάνετε τώρα ως Επίτροπος για την ενίσχυση αυτού του προγράμματος. Uh, certainly during the course of my time as minister in Εγώ προσπάθησα να μειώσω γενικότερα τις ε, γραφειοκροτικές επιβαρύνσεις. Ξέρω και ότι υπάρχουν περαιτέρω προβλήματα για τις ε, νησιωτικές περιοχές. Υπάρχουν ξεχωριστά προγράμματα για τις νησιωτικές περιοχές και κάποια επιμέρους προβλήματα ε, θα τα εξετάσουμε εφόσον μπορεί να επιληθούν και για τις απότερες περιφερειακές περιοχές και για τα νησιά. Τώρα το πρόβλημα το συγκεκριμένο στο οποίο αναφερθήκατε φυσικά δεν το γνωρίζω αλλά ίσως θα πρέπει να το συζητήσουμε για να βρεθεί μια λύση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σμιθ. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας καλωσορίζω Φιλ. Εγώ σαν Σκότος θαυμάζω, σαν Σκοτσέζο συγγνώμη, <laughs> θαυμάζω την Ιρλανδική Γεωργία και περιμένω αρκετά από την επόμενη πενταετία να δούμε ε, ποιο ουίσκι είναι καλύτερο, εγώ θα φέρω το δικό μας, εσείς το δικό σας και θα ε, διαγωνιστούμε. Και νομίζω ότι θα πάρουν πολύ μέρος στο διαγωνισμό αυτό. Επίσης ε, τα όσα είπατε ε, για ε, τα αμνοερήφια έχει μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε και να απλοποιήσουμε την κατάσταση χωρίς να χάσουμε τις, τα ωφέλη της ανιχνευσιμότητας. Τώρα σχετικά με τις τιμές που επιβάλλουν τα σούπερ μάρκετς νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είπατε να πάρει κάποια μέτρα για να υπάρξει μια πιο δίκαιη διαδικασία. Τι ακριβώς θέλετε να κάνετε, σκοπεύετε να κάνετε, γιατί υπάρχουν προβλήματα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας σχετικά με το ουίσκι. Έχω ταξιδέψει πάρα πολύ στη Σκοτία από το Όμπαν μέχρι την δυτική πλευρά και έχω συναντήσει πάρα πολλούς παραγωγούς. Και φυσικά το εκμεταλλεύτηκα όπως φαντάζεστε τώρα. Πράγματι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες σε σχέση με τον τελικό καταναλωτή και τα εμπορικά περιθώρια τα οποία θα έπρεπε σε ένα μεγαλύτερο βαθμό να πηγαίνουν στον παραγωγό. Έχει υπάρξει μείωση ε, του ποσοστού που πηγαίνει στον παραγωγό τα τελευταία χρόνια. Και γι' αυτό η συγκέντρωση της ενίσχυσης της αγοράς στα πλαίσια της αλυσίδας εμπορίας και στα σούπερ μάρκετ αυτή η υπερσυγκέντρωση έχει ενισχύσει την θέση τους αλλά ε, δεν έχει ενισχύσει την θέση των γεωργών. Υπάρχουν όμως κάποια προγράμματα τοπικά εθελοντικά και στη δική σας χώρα μέσω ε, διαπραγματεύσεων συλλογικών έτσι ώστε να υπάρξει πιο δίκαιη κατανομή του ποσοστού κέρδους και στα οποροκυπευτικά. Νομίζω ότι οι εθελοντικές δραστηριότητες ε, είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να διαχειριστεί κανείς και εξαρτάται από την καλή θέληση αυτών που συμμετέχουν στην διαδικασία στην αλυσίδα. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει στην παρούσα φάση μια πτώση της εμπιστοσύνη ανάμεσα στους παραγωγούς από τη μία και στα σούπερ μάρκετ από την άλλη. Και θα δούμε κάποιες νομοθετικές τροπολογίες στον τομέα των συγκεκριμένων εφόσον πράγματι από ό,τι φαίνεται υπάρχει κάποια δυσθυμία για την υπερσυγκέντρωση κάποιων επιχειρήσεων στον τομέα των τροφίμων πάντα. Ήρθε η ώρα του κύριου Άγνιου. Υπάρχει αντίφαση στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠΣ ό,τι αφορά τη ζάχαρη. Η βιομηχανία ζαχαροτέφλων θα απελευθερωθεί από τις ποσοστώσεις, ενώ για το ζαχαροκάλαμα δεν ισχύει το ίδιο. 200 θέσεις επηρεάζονται στην εκλογική μου περιφέρεια. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι... Ε, θα διορθωθεί η κατάσταση. Βέβαια, ε, τα εργοστάσια ζάχαρης δεν βρίσκονται μακριά από την αγορά. Και μήπως έτσι με, τις, ε, με, τα, νέα αυτά, με τα νέα αυτά μέτρα διακυβεύσουμε τη βιομηχανία. Πολλοί πια δεν θα μπορέσουν να, να καλλιεργήσουν κράβη και αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα. Συμφωνείτε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, έχουν τη διακριτική ευχαίρεια και να αποφασίζουν αν θα επιτρέψουν την ε, καλλιέργεια γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών. Ο κανόνας των τριών καλλιεργειών είναι κάτι το οποίο ε, μπορεί να δημιουργήσει περιθώρια καλής οργάνωσης και αύξησης κερδών. Θα δούμε σε ποιο βαθμό η πρακτική εφαρμογή θα δώσει αποδείξεις και στα πλαίσια της αναθεώρησης θα το εξετάσουμε. Αλλά η διαφοροποίηση των καλλιεργιών είναι βασικό συστατικό. Η πρακτική εφαρμογή ίσως να είναι δύσκολη, ανάλογα με το μέγεθος της εκμετάλλευσης, το είδος κτλ. Σχετικά τώρα με τη ζάχαρη. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα που είχε κάποτε βιομηχανία ζάχαρης και θα ήθελε να έχει πάλι στο μέλλον αρκεί να είμαστε αρκετά ανταγωνιστικοί. Βλέπετε ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί εδώ και σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία καμία βιομηχανία, οικονομική δραστηριότητα δεν την χάνει εγγυήσεων και ξέρουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με την παραγωγή ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ιδιαίτερα μετά το τέλος των ποσοστώσεων άνοιξαν πάρα πολλοί αγορές για τις τρίτες χώρες και αυτό έφυξε τις ε, περιοχές ε, ε, με τα ζαχαρότευτλα αλλά που είχαν και άλλα πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες μορφές παραγωγής. Όταν έρθω στην περιοχή σας όπως είπαμε θα τα επανεξετάσουμε όλα αυτά και να δούμε ακριβώς τι επιπτώσεις έχει η εφαρμογή του συγκεκριμένου κανόνα. Ίσως λοιπόν σύντομα να σας επισκεφθώ. Τώρα, σαν Υπουργός Περιβάλλοντος είχα ασχοληθεί με τα θέματα των γενετικά τροποποιημένων και στα πλαίσια των, της εξέτασης του θέματος από τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ. Εδώ φαίνεται ότι το θέμα της επικουρικότητας σε σχέση με την αδειοδότηση της καλλιέργειας αυτής είναι κάτι το οποίο είναι σε εκκρεμότητα. Ο κύριος Γιούνκερ είπε ότι αν τα κράτη-μέλη είναι κατά αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όπως επίσης και οι επιστημονικές σύμβουλες. Ε, το θέμα είναι ακόμα στην αρχή. Ευχαριστώ κύριε Σταντά. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, έχουμε διεθνείς διαπραγματεύσεις που θίγουν ε, τα γεωργικά μας προϊόντα. Οπότε οι γεωργοί μας ε, ανησυχούν πολύ. Αλλά και οι καταναλωτές που πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στην δηλωμένη ποιότητα των γεωργικών προϊόντων. Η, η υγειονομική ποιότητα των τρίτων χωρών, των προϊόντων των τρίτων χωρών πρέπει να είναι ίδια με αυτή που απαιτούμε από τα δικά μας προϊόντα. Και η παρουσία ορισμένων τομέων όπως της ε, ζάχαρης και του βοήου κρέατος πώς θα διατηρηθεί, πώς θα εγγυηθείτε την προστασία των προϊόντων μας και ότι θα διατεθούν στα πλαίσια δίκαιου ανταγωνισμού όταν καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις αυτές. Επαναλαμβάνω την ερώτηση που έκανε ο συνάδελφο Άντριου διαπραγματεύσεις αλικάν για τα ονόματα των κτημάτων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για πολλά προϊόντα μας. Βεβαίως, στα πλαίσια της ε, διαπραγμάτευσης για τις ε, γεωγραφικές ενδείξεις και το θέμα των κτημάτων. Ξέρω ότι αυτά ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και τους Γάλλους και άλλους στην Νότια Ευρώπη. Οι διαπραγματευτές μας το θεωρούν πολύ λεπτό θέμα και το έχουν υπόψη. Δεύτερον, όπως είπε και ο πρόεδρος Γιούνκερ, δεν θα θυσιάσουμε τη γεωργία μας για να σεβαστούμε προδιαγραφές. Υπάρχουν ευαίσθητοι τομείς όπως το βόιο, το ρύζι, τα πουλερικά που πρέπει να επιδιώξουμε να προστατεύσουμε γιατί χρειάζονται. Σίγουρα λοιπόν ε, δεν θα ειστερήσουμε ε, στην ανάγκη ενδεχομένω εισαγωγικών δασμών για να προστατεύσουμε τα προϊόντα. Οι προδιαγραφές είναι θέμα της Γενικής Διεύθυνσης ΣΑΝΚΟ αλλά από πλευράς γεωργίας οποιαδήποτε συμφωνία που έχουμε μέσω του TTIP για παράδειγμα με τις ΗΠΑ θα πρέπει να λάβει υπόψη τις προδιαγραφές. Δεν θα θυσιάσουμε το υψηλό επίπεδο προδιαγραφών που όλοι επιδιώκουμε να τηρούμε και που έχουμε όλοι αναπτύξει από τότε που είχαμε το πρόβλημα με την ασθένεια των βοηδών. Δεν θα τα θυσιάσουμε όλα αυτά μόνο και μόνο για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Η συμφωνία πρέπει να είναι ούτω ή άλλω σφαιρική, όχι μόνο σε θέματα γεωργίας. Ευχαριστώ. Πολύ χαιρόμαστε με αυτές τις διαβεβαιώσεις ο κύριος Ταραμπέλα. Κύριε Επίτροπε, κύριε Προτινόμενο Επίτροπε. Πρόσφατα ανέλαβα την έκθεση για το πρόγραμμα προώθησης ε, το, της κατανάλωσης απορροκυπευτικό και γάλακτος στα σχολεία. Τον Ιανουάριο του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διάλεξε το άρθρο 43.2 ε, ως νομική βάση με τη διαδικασία συναπόφαση. Το Συμβούλιο όμως φαίνεται και μάλιστα ομόφωνα σχεδόν ότι η νομική βάση θα πρέπει να είναι η παράγραφος 3 του 43, κάτι που αποκλείει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη διαδικασία λήψη αποφάσεων, κάτι που είναι απαράδεκτο με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνα. Δύο ερωτήσεις. Πέραν τη αθαρρυντική απάντηση που δώσατε, ε, θα μα διαβεβαιώσετε ότι θα προασπίσετε τα προνόμια και τι εξουσίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέχρι το τέλος τη διαδικασία ω προ τη συναπόφαση και φυσικά θα διαφυλάξετε και τον προϋπολογισμό. Τώρα, δεν θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εντάξει αυτό το πρόγραμμα σε, ένα, σε μια ευρύτερη προσπάθεια καλ, καλύτερης διαπαιδαγώγησης για την υγιεινή διατροφή. Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Σας ευχαριστώ. Φυσικά. Είμαι υπέρα του άρθρου 43. Αυτή είναι η ενδεδειγμένη νομική βάση και η συναπόφαση για το καθεστώς ε, για την ένταξη των απορροκυπευτικών και του γάλακτος στα σχολεία. Και μάλιστα το καθεστώς αυτό ε, δεν ε, αναφέρεται μόνο στα νοπά απορροκυπευτικά αλλά και στα μεταποιημένα και στους χυμούς φρούτων. Και η νέα πρόταση για τα σχολεία από τον Ιανουάριο του 2014 μιλά για την διανομή ε, στα σχολεία, κυρίως ε, νοπών απορροκυπευτικών και γάλακτος. Και χαίρομαι που αναλάβατε την έκθεση. Θυμάμαι στα μέσα Σεπτεμβρίου στην Ολομέλεια συζητήθηκε το θέμα αυτό και χαίρομαι που αναλάβατε εσείς την σχετική έκθεση. Οπότε περιμένουμε ανυπομονησία την πρόταση που θα υποβάλλετε για το συγκεκριμένο αυτό θέμα και για τα ειδικά μέτρα διανομής στα σχολεία απορροκυπευτικών και γάλακτος και να... θα δούμε πώς θα το προωθήσουμε. Πάντως σας διαβεβαιώ ότι θα υποστηρίξω την νομική βάση του 43.2. Ο κύριος ε, ευχαριστώ. Κύριε Χόγκεν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι για τις εξαιρέσεις για τους κτηνοτρόφους. Η οδηγία για τις βιοάδειες. Δίνει δυνατότητα να υπάρξει πατέντα για κάποια φυτά. Όμως ε, οι κτηνοτρόφοι πάντα είχαν δυνατότητα να αναπτύξουν και να διαθέσουν νέα είδη χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουν ε, τεράστια ποσά σε αυτούς που έχουν τις πατέντες ε, Θεωρείτε λοιπόν ότι πρέπει να διατηρηθεί αυτή η εξαίρεση για τους κτηνοτρόφους, ούτως ώστε οι μικροί κτηνοτρόφοι να μπορούν να αναπτύσσουν νέα είδη. Θα το υπερασπιστείτε αυτό έναντι του συναδέλφου σας που έχει το χαρτοφυλάκιο για την εσωτερική αγορά. Ο τομέας αυτός είναι πολύ καινοτόμο στην Ιρλανδία και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό για μας αυτό. Έχω υπόψη μου την έκθεση για τη δημιουργία νέων ε, φυτών της κυρίας Πόλσεν για αυτό το τομέα. Η έκθεση αυτή είναι πολύ σημαντική για να μπορούμε να θρέψουμε τον πληθυσμό μας ε, σε μεταβαλλόμενο κλίμα και είναι πολύ σημαντικός για τους κτηνοτρόφους. Αλλά δεν μπορώ να δεσμευθώ ότι θα σας υποστηρίξω για αυτό που είπατε. Είναι κάτι που πρέπει να συζητήσω με τον Επίτροπο για την Εσωτερική Αγορά και θα το κάνω αυτό. Αλλά δεν μπορώ να δεσμευθώ σήμερα ε, Μία καλή συμβουλή που μου δώσανε πριν έρθω σε αυτήν την επιτροπή ήταν ότι μη δώσετε υποσχέσεις που δεν θα μπορούσατε να τηρήσετε. Θα το εξετάσω το θέμα αυτό. Έχω υπόψη μου τη σημασία που έχει η εξέλιξη νέων ειδών στη χώρα σας. Και λαμβάνω υπόψη μου τις προτάσεις που έκανε η καλή μας φίλη κυρία Πόλσεν. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Πάουλσεν αναφέρθηκε το όνομά της, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα κάνω μια διαφορετική ερώτηση. Δεν θα μιλήσω για την επιλογή των νέων ειδών, εν αλλά υπάρχει μια ευκαιρία νομίζω για τους Ευρωπαίους γεωργούς στην παρούσα φάση. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, οι οποίοι όμως εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο και ακριβώς αυτό ε, διευρύνει τις δυνατότητες ερμηνείας και δημιουργεί σύγχυση και για ε, το, την εκτροφή χείρων και για άλλα ζώα οι έλεγχοι και οι κανόνες εφαρμόζονται με διαφορετικό τρόπο. Το ίδιο και για τη μεταφορά των ζώων. Επίσης υπάρχουν διαφορετικοί τύποι εφαρμογής των κοινοτικών ρυθμίσεων. Ε, αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται με ομοιογενή τρόπο για όλους τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Έτσι δεν είναι. Στηρίζεται την ιδέα αυτή και θα πρέπει επίσης και να στηριχθεί η άποψη που εκφράζει το Κοινοβούλιο έτσι ώστε να υπάρξει μια νέα διαφορετική νομοθετική ρύθμιση. Έχω την αίσθηση ότι την τελευταία δεκαετία σε σχέση με την ευημερία των ζώων έχει υπάρξει πρόοδος και η παραγωγή είναι πιο ικανοποιημένη γιατί ξέρετε ότι παλιότερα υπήρχε ε, διαφορετική άποψη ενώ τώρα θεωρείται ότι ένα ευτυχές ζώο είναι ένα ζώο καλό για την κατανάλωση. Λοιπόν, ε, ε, ε, ξέρω τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν τους κανόνες οι Σουηδοί σε σχέση με την ευημερία των ζώων. Γνωρίζω λοιπόν αυτό το οποίο θίξατε σαν θέμα και θα ήθελα πράγματι να το συζητήσω μαζί σας να υπάρξει περαιτέρω εναρμόνιση ε, σε σχέση με το θέμα των Σουηδών το οποίο μου το θέσατε και ιδιωτικά. Υπάρχει βέβαια μια δυσκολία, δεν είμαι επίτροπος ακόμα, αλλά αν γίνω επίτροπος στο μέλλον σίγουρα το θέμα αυτό θέλω να το συζητήσω εκ νέου μαζί σας για να πετύχουμε καλύτερη ε, και πιο ομοιογενή εφαρμογή των μέτρων που στοχεύουν στην ευμερία των ζώων. Ευχαριστώ πολύ. Αρχίσουμε τον κύριο Μπούντα τώρα ε, ε, για τον επόμενο γύρο ομιλητών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιο Επίτροπε, το 2012-2013 είχαμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην ε, νομοθεσία για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Προσαρμογή λοιπόν στις νέες συνθήκες. Όμως η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ δεν έλυσε το πρόβλημα των μεγάλων διαφορών μεταξύ αμέσων πληρωμών που δίνονται σε διάφορα κράτη-μέλη και τις πληρωμές που λαμβάνουν οι γεωργοί στις ε, χώρες Ανατολικής Ευρώπης. Οι τελευταίες αυτές πληρωμές ήταν πολύ χαμηλότερες. Το νομοθετικό πακέτο που άρχισε να ισχύει το 2013 καθορίζει ότι οι πληρωμές αυτές θα έπρεπε να είναι ψηλότερες. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μεγάλη ανισότητα και αυτό οδηγεί και σε ανισότητα μεταξύ γεωργών. Και επειδή υπάρχουν τώρα νέες προκλήσεις λόγω του ρωσικού εμπάργου, θέλω να ρωτήσω συγκεκριμένα εάν θα τροποποιήσετε το χρονοδιάγραμμα για την αύξηση των πληρωμών προς, το, προς τα κράτη-μέλη και αν προβλέπετε και άλλα μέτρα στήριξης για τους παραγωγούς σε κάποια κράτη-μέλη για να καλυφθούν αυτές τις διαφορές. Ευχαριστώ πολύ. Φαντάζομαι ότι δεν μπορούμε ως διαμαγείας να λύσουμε το πρόβλημα. Και αυτό θα το διαπιστώσατε και στην Επιτροπή σας. Γιατί υπάρχει διάσταση απόψε μεταξύ των κρατών μελών για το ρυθμό και το εύρος ε, της εξωτερικής αυτής σύγκλησης. Πάντως χώρες όπως η Εστονία, Λιθουανία, Λετωνία έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στη σύγκληση. Και τέθηκε ένα νότο το όριο στο μέγιστο ποσοστό άμεσων ενισχύσεων και αυτό δεν ήταν εύκολο για τις χώρες ε, που έχουν μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις να το δεχτούν, αλλά πέρασε τελικά και στα μέτρα που θεσπίστηκαν έγιναν προσπάθειες και σημειώθηκε πρόοδος για τις χώρες που είχαν χαμηλότερο επίπεδο πληρωμών. Θα δούμε τελικά πώς θα εφαρμοστούν τα μέτρα που εγκρίθηκαν και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την ελαστικότητα που δώσαμε στα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη μπορούν να, να θεσπίσουν και επιπλέον μέτρα για να επιτύχουν αυτή τη σύγκληση στο εσωτερικό τους. Και με τα στοιχεία που θα συγκεντρώσουμε θα προβούμε στην ενδιάμεση αναθεώρηση και θα δούμε κατά πόσο υλοποιήσαμε τους στόχους ε, της ΚΑΠ. 8.000 τροπολογίες κατατέθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ΚΑΠ τεράστιο έργο, αξιοσημείωτη προσπάθεια και θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία. Φαίνεται από τις στατιστικές πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουμε ότι κάποια πρόοδο σημειώθηκε. Βέβαια, ποιο είναι το επίπεδο της πρόοδου, για αυτό το θέμα δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Νόιντσολ. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, Θέλω να σας μιλήσω από πλευράς της Ευρωπαϊκής Μελισσοκομείας. Η μελισσοκομεία είναι σημαντικότατη δραστηριότητα. Επιπλέον, οι μέλισσες είναι ένδειξη για την υγεία της ε, υπαίθρου. Οι μέλισσες θέτουν τις ε, τρεις ερωτήσεις. Θα δώσετε προτεραιότητα στην ε, διατήρηση της, όλων των ειδών των μελισσών. Επιπλέον, θα αποφύγετε τη χρήση νέων νοικοτινοειδών που δημιουργούν προβλήματα στην επιβίωση. Επίσης, θέλουμε οι μέλισσες να μην ε, χρειαστεί να ε, ζουν σε συνθήκες ε, σε συνθήκες τροποποιημένο, γενικά τροποποιημένων καλλιεργιών γιατί οι μέλισσες δεν γνωρίζουν σύνορα και μπορεί να πάνε και σε αυτές. Όπως ξέρετε εδώ και πολλά χρόνια, η κοινή γεωργική πολιτική έχει στηρίξει τον τομέα της μελισσοκομείας μέσω των εθνικών ε, μελισσοκομικών ε, προγραμμάτων και ε, στηρίζουμε την παραγωγή μελιού. Τα γράμματα για το 2016, μέχρι το 2016 ισχύουν στα κράτη-μέλη και τα τελευταία χρόνια, από ό,τι καταλαβαίνω, η Κομισιόν πήρε μέτρα για να ε, κάνει πιο αυστηρή την ε, έγκριση των ε, παρασιτοκτόνων. Οι νέοι κανόνες για τη μείωση των επιπτώσεων από τα παρασιτοκτόνα στο περιβάλλον και τον άνθρωπο έχουν εισαχθεί και κάνουμε χρήση και μη χημικών μεθόδων και χαμηλή χρήση παρασιτοκτόνων. Έτσι συμπληρώνουμε τα μέτρα που προβλέπονται γενικά στην κοινή γεωρική πολιτική για να προωθήσουμε τη βιοπικιλότητα. Τώρα για τα θέματα ε, της απαγόρευσης των ε, νέων κοτινοειδών είναι θέμα σάνκο, αλλά έχουν γίνει μελέτες που λένε ότι κάποια τέτοια προϊόντα είναι τεράστιος κίνδυνος για τις μέλισσες και γι' αυτό έχουμε περιορίσει πάρα πολύ τη χρήση τους σε ορισμένους τομείς και σε δύο χρόνια θα δούμε εκ νέου τις συνθήκες για τη χρήση τους με βάση τις ε, νέες επιστημονικές γνώσεις και φυσικά θα ενημερώσω την Επιτροπή για τι μέτρα θα λάβουμε. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Πετήρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Χόγκαν, όλο και περισσότεροι άνθρωποι, κυρίως νέοι, αφήνουν ε, ε, την Ήπεθρο και πηγαίνουν στα, στις μεγάλες πόλεις ε, για να επιβιώσουν. Θα πρέπει όμως να κρατήσουμε την Ήπεθρο ζωντανή και γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε συνθήκες ε, και φυσικά καλύτερη οικονομική, κοινωνική και δημοτική υποδομή και φυσικά κάποιες πηγές εισοδήματος. Τι μέτρα θα αναλάβετε προκειμένου να δώσετε ενάψματα για την παραμονή των αγροτών μας και του αγροτικού πληθυσμού στην Ήπεθρο. Γιατί στην Ήπεθρο παράγουμε τρόφιμα, στην Ήπεθρο διαφυλάσσουμε την βιοποικιλότητα. Οι αγρότες μας είναι και του περιβάλλοντος. Με ενδιαφέρει λοιπόν αν αναλάβετε το χαρτοφυλάκιο της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης θα προτείνετε κάποια μέτρα για την σωστή αμοιβή, για τη φύλαξη του χώρου και του περιβάλλοντος. Υπάρχουν. Ε, Ότι ήδη υπάρχει μεγάλη υποστήριξη για, από τις άμεσες ενισχύσεις στο θέμα του πρασινίσματος και της αγροτικής ανάπτυξης. 40% των κονδυλίων θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν περιβαλλοντικά μέτρα στην Ήπεθρο, στις αγροτικές περιοχές. Και υπάρχουν ήδη μέτρα της κοινή γεωργικής πολιτικής για να ε, υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι. Επιπλέον, στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και με το Leader δίνουμε δυνατότητες για οικονομική ανάπτυξη, για κοινωνικό κεφάλαιο, για στοιχειώδεις υπηρεσίες και για ειδικά μέτρα που είναι σημαντικά για την διαφύλαξη της υπαίθρου. Και όλες οι χώρες έχουν υποβάλει σχέδια δράσης, πολλοί άριθμα έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να εξεταστούν και να δούμε κατά πόσο τηρούνται οι στόχοι ανάπτυξη πέθρου. Το θέμα είναι πώς οι νέοι και ο αγροτικός πληθυσμός που δεν ε, έχουν ε, μεγάλη επαγγελματική δραστηριότητα να μπορούν να εξασφαλίσουν συγχρηματοδότηση για πολλά από τα μέτρα που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στραφούμε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και σε διάφορους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για να εξασφαλίσουμε περαιτέρω κονδύλια στα πλαίσια της χρηματοδότησης για να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα στην Ήπεθρο, περισσότερες θέσεις απασχόλησης και μεγαλύτερη βιωσιμότητα και ζωτικότητα της Ήπεθρο. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Σας ευχαριστώ. Μερικοί θεωρούν ότι η κοινή αγροτική πολιτική θα πρέπει να χαρακτηριστεί κοινή γεωργική και περιβαλλοντική πολιτική. Ευχαριστώ. Φτάνουμε στο τέλος κύριε Χόγκαν. Κουράγιο. Άκουσα με ευχαρίστηση αυτό που είπατε για την σημασία που έχει η μείωση της εκπομπής καυσαερίων. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα όπως επίσης και την ε, διάβρωση των ανωτέρων στρωμάτων του εδάφους. Ε, εσείς πιστεύετε ότι οι κανόνες για την προστασία της ε, γης εφαρμόζονται σωστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή πιστεύετε ότι απειλείται η ανθεκτικότητα της, ε, των ε, γεωργικών καλλιεργειών. Πράγματι έχουν υπάρξει αρκετά μέτρα και αρκετές πιστώσεις και στα πλαίσια των διαδικασιών πολλαπλής συμμόρφωσης γύρω από τα θέματα αυτά, τα οποία γνωρίζω επειδή ασχολήθηκα ιδιαίτερα και με την οδηγία για την ποιότητα των υδάτων ενδιαφέρθηκα για την κοινή αγροτική πολιτική και παρακολούθησα αυτά τα οποία έχετε προτείνει έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των ε, εδαφών και των υδάτινων πόρων στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρησιμοποιούνται για γεωργική παραγωγή και για παραγωγή τροφίμων. Υπάρχουν προβλήματα λοιπόν σε πολύ μεγάλα ποσοστά, άνω του 40% των εδαφών. Ε, μέτρα έχουν προταθεί, ε, αλλά υπήρχαν και διαφωνίες φυσικά ακριβώς για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε ε, τις πηγές των υδάτινων πόρων και να ελέγξουμε την ποιότητά τους. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στον επόμενο γύρο, τον 8ο. Η κυρία Εράντς Γκαρσία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε υποψήφιο επίτροπε, με ιδιαίτερη χαρά σας άκουσα να λέτε για βελτίωση της αλυσίδας ε, τροφίμων. Άλλωστε η σχετική ισπανική νομοθεσία έχει αποφέρει καρπούς. Τα προκυπευτικά είναι τα μεγάλα θύματα της ε, αλυσίδας τροφίμων. Θα προτείνετε μια πλούστευση για το 2015, είπατε. Αντί για πλούστευση θα προτιμούσα βελτίωση. Γιατί το καθεστώς για τα απορροκυπευτικά δεν έχει καλό σύστημα διαχείρισης των κρίσεων. Θα υποβάλλετε και σκέλος διαχείρισης κρίσεων στην πρότασή σας για τα απορροκυπευτικά. Δεύτερη ερώτηση. Ο κανονισμός ε, ΠΟΣΕΙ για τις ε, άκρος απόκεντρες περιοχές δεν αναφέρθηκε καθόλου. Πολύ σημαντικό πρόγραμμα αυτό για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Μάλιστα ε, η προηγούμενη πρόταση δυστυχώς βάγισε. Θα υποβάλλετε νέα πρόταση για το καθεστώς ΠΟΣΕΙ, το καθεστώς δηλαδή για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Ευχαριστώ. I Όντως, υπήρχε πολιτική για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές με βάση το πρόγραμμα ΠΟΣΕΙ πολύ σημαντικό πρόγραμμα και καθεστώς. Κατοχυρώθηκε από τις συνθήκες πριν από πολλά χρόνια και αφορούσε ιδιαίτερα τα νησιά. Εκρεμεί αναθεώρηση του ΠΟΣΕΙ και θα σας ενημερώσω για την πορεία της το 2015. Ήδη έχουμε ένα πρόγραμμα για την Πορτογαλία για τη στήριξη της γαλακτοπαραγωγής. Λαμβάνουμε υπόψη το ενεργειακό κόστος, το κόστος μεταφοράς και το επιπλέον κόστος που αναλαμβάνουν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές ε, όταν πρέπει να φέρουν προϊόντα τους προς την υπηρετική Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά την διαχείριση των κρίσεων, έχουμε ολόκληρη εργαλειοθήκη με μέτρα αγοράς για την κρίση. Έχουμε μέτρα παρέμβασης, ιδιωτικής αποθήκευσης, και εξαγωγικές επιστροφές. Όλα αυτά είναι μέτρα αγοράς για τη διαχείριση κρίσεων σε ευαίσθητους τομείς. Και εξαιτία της γεωπολιτικής κρίσης που δημιουργήθηκε μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Όλα αυτά τα μέτρα θα τα χρησιμοποιήσουμε στο έπακρο. Και ο Επίτροπος Τσόλος εξήγηλε ήδη συμπληρωματική ενίσχυση Βέβαια έχει προβλήματα με τη Γενική Διεύθυνση Προπολογισμών για να εξασφαλίσει αυτά τα συμπληρωματικά κονδύλια. Θέλουμε ισορροπημένο προπολογισμό αφενό, αφετέρου να βρούμε είτε στο αποθεματικό μα είτε στα περιθώρια που έχουμε επιπλέον κονδύλια για να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των γεωργών μα των παραγωγών μα. Αυτό που ενδιαφέρει και εσά, δηλαδή. Σα ευχαριστώ. Ο κύριο Ρεμπέγκα. Ε, Ευχαριστώ κύριε υποψήφιε για αυτά τα οποία μας είπατε. Ε, τέθηκε το θέμα των νέων αγορών για τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της έβρωσης νέων αγορών. Και αυτό προκλήθηκε σημαντικό πρόβλημα γύρω από αυτό μετά από το εμπάργο με τη Ρωσία. Για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την παγίδα στην οποία έχουμε πέσει χωρίς να δημιουργούμε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που θα έχουν έτσι και αλλιώς και περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις στις αγορές και στις καταναλωτές ε, πρέπει να πάρουμε μέτρα τα οποία ε, υποστηρίζουν βέβαια ε, τη δημιουργία των θέσεων απασχόλησης αλλά μόνο θεωρητικά εσείς θα προβλέψετε κάποια οικονομική βοήθεια για την αύξηση των εξαγωγών και πότε θα πάρετε τα κατάλληλα μέτρα ή θα περιμένουμε ένα χρόνο πρώτα. Οι παραγωγοί δεν μπορούν να περιμένουν. Δέχομαι το ότι οι παραγωγοί πράγματι δεν είναι σε θέση να περιμένουν και βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δράσει όμως με ταχύτητα. Ήδη από τον μήνα Αύγουστο και ο Επίτροπος Τσίολος ε, προσπαθεί έτσι ώστε αν χρειαστεί να ληφθούν και περαιτέρω μέτρα. Ήδη ανακοίνωσε τα 168 εκατομμύρια, τώρα το πώς θα συγκεντρηθούν τα χρήματα αυτά ε, είναι κάτι το οποίο είναι ακόμα προσυζήτηση, αλλά είναι κάτι που θα γίνει πάντως. Εγώ είπα επίσης ότι υπάρχει μια βελτιωμένη πρόταση από το 15 και μετά για την προώθηση των εξαγωγών αντί για 60 εκατομμύρια στην προηγούμενη περίοδο θα υπάρξουν 200 για αυτήν την προγραμματική περίοδο. Αυτό θα μας βοηθήσει να ανοίξουμε νέες προοπτικές αγορών και θα μειώσει τις πιέσεις οι οποίες, οι οποίες υφίστανται στις δύσκολες γεωγραφικά αγορές σήμερα. Νομίζω ότι όλα αυτά τα θέματα και όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και μέσω των πρέσβεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως λέμε και μέσω των προγραμμάτων βοήθειας προς άλλες χώρες θα μας βοηθήσουν να μειώσουμε την εξάρτηση που έχουμε από διάφορες περιοχές γεωγραφικά ευαίσθητες πολιτικά σήμερα. Ε, εμείς τα μέτρα αυτά θα προσπαθήσουμε ε, να τα περάσουμε και στα πλαίσια του συνόλου των επιτρόπων θα δούμε τι μας δίνει και ο προϋπολογισμός και έτσι θα γνωρίζουμε πόσο γρήγορα θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των παραγωγών. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μέλο. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, ελπίζω να αναλάβετε καθήκοντά σας και έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Τι γίνεται με την ανανέωση των γενεών στη Γεωργία, γιατί δεν θα έχει μέλλον η Γεωργία αν δεν προσελκύσουμε νέους αυτή. Και στατιστικά ένας γεωργός, ε, ε είναι, ε, ένας στους εννέα γεωργούς μόνο είναι κάτω των 35 ετών. Πολύ ανησυχητική ε, αυτή η πληροφορία για την Ισπανία, Πορτογαλία, Βουλγαρία. Ε, που έχουν ακόμη χειρότερη κατάσταση. Ένας μόνο νέο κάτω 35 για 25, για 20 συγγνώμη. Ενώ η Πολωνία, η Αυστρία ε, έχουν ένα νέο γεωργό για τρει ε, άνω των 55 ετών γεωργούς. Μεγάλη διαφορά δηλαδή μεταξύ των κρατών μελών για την ανανέωση της γεωργίας και την προσέλκυση νέων. Βλέπετε τι τεράστιες διαφορές υπάρχουν τι προτείνετε να κάνετε για να προωθήσετε αυτή την ανανέωση, την αναγέννηση της γεωργίας και φυσικά χρειάζονται επιπλέον πόροι για την ανανέωση αυτή των γενεών στη γεωργία. Ξέρω βέβαια ότι ε, έχουμε πίεση και συρρήκνωση του γεωργικού μας προϋπολογισμού. Ποια θα είναι η δική σας θέση, θα προτείνετε αύξηση ή συρρήκνωση του γεωργικού προϋπολογισμού και της μεταρρύθμισης ΚΑΠ κάνω ό,τι μπορώ για να διατηρηθεί ο προπολογισμό. Και πιστεύω ότι μπορούμε να μοχλέψουμε από τους τομείς άλλων επιτρόπων ε, χρηματοδοτήσεις μέσω του ορίζον 2020 και σε άλλους τομείς και από άλλους τομείς και θα προσπαθήσω να αξιοποιήσω και όλες τις δυνατότητες που έχουμε για δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ήπεθρο ούτω ώστε όσοι έχουν ε, δυσχέρει αυτή τη στιγμή λόγω τη οικονομικής χρήση να πάρουν δάνεια από τράπεζες, να λάβουν χρηματοδοτήσει. Αυτά είναι πραγματικά θέματα για πραγματικούς ανθρώπους και, πραγματικά, και ιδίως τους νέους. που δεν έχουν εύκολα πρόσβαση στις τράπεζες. Και οι ανανεώσιμες βοηθάει. Βοηθάνε και ιδίως βοηθάνε στις ε, διαθροτικές μεταρρυθμίσεις που χρειαζόμαστε. Το γεγονός ότι 69% των εκμεταλλεύσεων είναι μικρές και πολλές από αυτές είναι εκμεταλλεύσεις ε, που τις τρέχουν γυρεότεροι ε, γεωργοί είναι ανισχυτικό. Πρέπει να δούμε πώς με εταιρικέ σχέσεις μεταξύ κρατών μελών. Ξέρετε, όταν δίνουμε πολλές ε, ενισχύσεις σε γυρεότερους γεωργούς, ε, πολλές φορές δεν τους ενθαρρύνει να συνταξιοδοτηθούν για να δώσουμε ευκαιρίες στους νέους. Πρέπει να δούμε. Πολλές, ε, πολλές φορές είναι και θέμα ότι οι γυρεότεροι φοβούνται ότι το εισόδημά τους θα πέσει πάρα πολύ αν βγουν από την παραγωγή. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε πόρους πέρα από το 25% επιπλέον επί του οποίου ε, επέμεινε το Κοινοβούλιο, ούτω ώστε να πάρουν οι νέοι γεωργοί χρηματοδοτήσει στα πλαίσια τη νέα ΚΚΠ. Σα ευχαριστώ κύριε Σκαπούτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον υποψήφιο Επίτροπο. Εγώ θα μιλήσω για κάτι το οποίο δεν συζητάμε συχνά στη Γεωργία, αλλά βασικό για την αηφόρο ανάπτυξη. Την έρευνα ε, και την καινοτομία. Η γεωργική ε, έρευνα στην Ευρώπη είναι πολύ διασπασμένη. Συνήθως οι πόροι πηγαίνουν στη βασική έρευνα και όχι στις εφαρμογές της σε επίπεδο επιχείρησης οι σχέσεις γεωργίας επιστήμης για τις νέες λύσεις και νέες εφευρέσεις και τα λοιπά σίγουρα θα πρέπει να καταστήσουν ε, ε, πιο πλούσια και πιο ανταγωνιστική τη γεωργία την ευρωπαϊκή και σε οικονομικό επίπεδο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Εσείς θα είσαστε υπεύθυνος για την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας και της καινοτομίας και στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Ποια είναι η γνώμη σας. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η μετάδοση των γνώσεων και η έρευνα και η καινοτομία θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα, ιδιαίτερα όταν έχουμε χαμηλά γεωργικά εισοδήματα. Νομίζω λοιπόν ότι και στα πλαίσια του προγράμματος για τις ε, κοινωνικές ε, προκλήσεις ε, είναι ιδιαίτερα υψηλό για τα επόμενα χρόνια που φτάνει uh, Φτάνει σε πάρα πολύ υψηλά ποσά και νομίζω ότι η κατανομή των χρημάτων αυτών θα μπορέσει να αποδώσει σε διάφορους τομείς. Και στα πλαίσια των προγραμμάτων για το 2020 θα βοηθήσουμε τους νέους και σε επίπεδο κατάρτισης έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι θα βρούμε τρόπους για να βοηθήσουμε τους νέους με νέες ιδέες, νέες πρωτοβουλίες, νέες μεθόδους ερευνητικές πώς θα παράγουμε περισσότερο μια εποχή που θα έχουμε λιγότερους σπόρους, που έχουμε λιγότερους σπόρους στη διάθεσή μας. Υπάρχουν μέτρα επίσης που περιλαμβάνονται και στα προγράμματα για την ανάπτυξη της υπαίθρου και εκεί υπάρχουν προτάσεις καινοτόμων εταιρικών σχέσεων ή μάλλον εταιρικών σχέσεων με στόχο την καινοτομία έτσι ώστε ε, τα προγράμματα αυτά να προωθηθούν και να τα προσφέρουμε στα κράτη-μέλη για να πετύχουμε τους στόχους τους οποίους σωστά έχετε υπογραμμίσει. Περνάμε στο δέκατο γύρο. Ο κύριος Έρντος, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Η αύξηση της αρδευόμενης ε, καλλιεργήσιμης γης είναι πολύ σημαντική. Στη Γεωργία, στην Ουγγαρία έχουμε παρικές είδωρ για άρδευση και το πρόγραμμα της γεωργίας ε, που στη χώρα μου θα βελτιώσει την κατάσταση. Θέλουμε όμως τη βοήθειά σας. Τρεις ερωτήσεις λοιπόν. Θεωρείτε ότι έχει μεγάλη σημασία η αύξηση της αρδευόμενης ε, καλλιεργούμενης γης. Δεύτερον, πέρα από την, ε, τους πόρους για την ανάπτυξη της υπαίθρου, της υπαίθρου τι πόρους μπορείτε να αξιοποιήσετε για να αναπτύξουμε νέα αρδευτικά συστήματα και τι θα κάνετε ούτω ώστε αυτά τα νέα αρδευτικά συστήματα να εφαρμοστούν στα πλαίσια των επενδύσεων για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Ε, νομίζω ότι η ερώτησή σας ε, τονίζει ακριβώς τη διαφορά μεταξύ Βόρειας και Νότιας Ευρώπης και τι πρέπει να κάνουμε, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε επαρκή ποσότητα και ποιότητα υδάτων για την ε, παραγωγή τροφίμων. Τα κράτη-μέλη για πρώτη φορά έχουν δυνατότητα να στηρίξουν επενδύσεις στην ε, άρδευση μέσω των προγραμμάτων επέκτασης της υπαίθρου. Έχουμε λοιπόν ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο για τους γεωργούς και για τις περιφέρειες στα πλαίσια του προγράμματος ανάπτυξης υπαίθρου για την άρδευση. Μπορούμε να στηρίξουμε λοιπόν τον εξοπλισμό στις εκμεταλλεύσεις για την άρδευση και τις εκτός εκμεταλλεύσεων υποδομές να βελτιώσουν τις υπάρχουσες υποδομές, να δημιουργήσουν νέες περιοχές όπου υπάρχει άρδευση. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις όμως αυτές μας επιτρέπουν να αποφύγουμε την αβεβαιότητα που υπήρχε και είναι ε, συμβατές με την οδηγία ε, πλαίσιο για τα ύδατα και θα μας επιτρέψουν να αξιοποιήσουμε πλήρως τις περιοχές όπου υπάρχει επαρκές νερό. Σε περιοχές λοιπόν που υπάρχουν προβλήματα, οι συνθήκες είναι πολύ πιο αυστηρές. Ελπίζω λοιπόν τα κράτη-μέλη θα έχουν την αναγκαία ευελιξία ούτω ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε και άλλες περιοχές ε, στην παραγωγή τροφίμων. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σάνι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε. Σήμερα το πρωί μιλήσαμε εκτελώς, εκτενώς για τη λειτουργία της κοινή γεωρικής πολιτικής. Δεν θα πρέπει όμως να μιλήσουμε και για τους στόχους της κοινή γεωρικής πολιτικής. Πιστεύω, όπως και άλλοι, ότι στόχος της κοινή γεωρικής πολιτικής είναι η παραγωγή ποιοτικών τροφίμων σε δίκαιες και προσιτές τιμές στην Ευρώπη. Θέλουμε τα τρόφιμα που φτάνουν στα τραπέζια των συμπολιτών μας, των 500 εκατομμυρίων συμπολιτών μας, να είναι υγιεινά και σε προσιτές τιμές. Δυστυχώς 100 εκατομμύρια συμπολίτες μας βρίσκονται στο όριο του υποσυτισμού. Και μάλιστα η κυβέρνησή μας έχει επιβάλει 20% φόρο στα τρόφιμα. Οπότε οι πιέσεις για, το θέμα, για τα τρόφιμα και η επιστηστική ασφάλεια είναι θέμα σημαντικό και έχει τεράστιες κοινωνικές διαστάσεις. Θα αναλάβετε την ευθύνη σας και τι μέτρα θα προτείνετε προκειμένου να τεθεί ένα τέρμα στον υποσυτισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εξασφαλίσουμε επιστημιστική ασφάλεια. ο πρώην Υπουργό Περιβάλλοντο στην Ιρλανδία, συμμετείχα στι διαπραγματεύσει για την κλιματική αλλαγή που είχαν στα πλαίσια της πλατφόρμας του Durban και το θέμα των τροφίμων και της επιστημιστική ασφάλειας. Άρα, σέβομαι πλήρω την ε, επιχειρηματολογία που στηρίζει την ερώτησή σας είναι τεράστιο θέμα που πολλοί στα πλαίσια της ζήτησης για τα τρόφιμα το αγνοούν. 870 εκατομμύρια στον πλανήτη μας πάσχουν από υποσυτισμό. Παρά το ότι υπάρχει επαρκής, υπάρχουν επαρκή τρόφιμα στον πλανήτη μας. Δεν μπορώ να παρέμβω τώρα στην ε, εθνική φορολογία, το ξέρετε αυτό. Είναι θέμα των πολιτικών προτεραιοτήτων των κρατών μελών. πολλά κράτη-μέλη δεν ε, έχουν καθόλου φόρους επί των τροφίμων. Δεν μπορώ να σχολιάσω την φορολογική ε, πολιτική των κρατών μελών, αλλά ο επισητισμός και τα τρόφιμα είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση σε νέες αγορές, που θα δώσει για την Ευρώπη περισσότερες ε, δυνατότητες εξαγωγών, ίσως με κάποια βοήθεια από πλευρά μας. Υπάρχουν θέματα που σχετίζονται με τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις. Θα κάνω όμως ό,τι μπορώ για να βοηθήσω την αρμόνιση, την απλούστευση, τη μείωση της γραφειοκρατίας για την παραγωγή τροφίμων και θα προστατεύσω και, τα δικαιώματα των καταναλωτών. Μάλιστα και περνάμε στον ενδέκατο γύρω ερωταπαντήσεων και δίνω το λόγο στον κύριο Καλινόφσκι. Σας ευχαριστώ. Πληθώρα ερωτήσεων. Πολλές αφορούσαν και το ρωσικό εμπάργο και την έλλειψη ανταγωνιστικότητας εξαιτία των άνισων πληρωμών. Πώς βλέπετε το μέλλον των βιοκαυσίμων τρίτης γενιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα βιοκαύσιμα υποτίθεται θα περιόριζαν τις εκπομπές καυσαερίων, κυρίως διοξιδίου του άνθρακα και θα ενίσχυαν το αγροτικό εισόδημα. Έχουμε όμως όλο και περισσότερα συστατικά βιοκαυσίμων ή έτοιμα τρίτα ε, βιοκαύσιμα που καταφθάνουν και κατακλείσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Τι γίνεται λοιπόν, τι γνώμη έχετε, πώς θα ληφθεί υπόψη η παραγωγή των ε, βιοκαυσίμων ε, σε ό,τι αφορά την έμεση αλλαγή χρήσης γης και θα υπάρχει διαφορά στα βιοκαύσιμα ανάλογα με το αν παράγονται με πρώτες ύλες ε, κοινοτικές ή με πρώτες ύλες προέλευσης τρίτων χωρών. Η συζήτηση για τα βιοκαύσιμα έχει αλλάξει πορεία, έχει πάρει διαφορετική στροφή τη τελευταία δεκαετία. Πριν από 10 χρόνια ήμασταν πολύ πιο ενθουσιώδεις για τα βιοκαύσιμα και τότε ήμουν μέλος της Ελλαδικής Βουλής και πράσινη έκαναν, ασκούσαν πιέσεις για την αύξηση το, της παραγωγής βιοκαυσίμων. Βέβαια, αναγνωρίστηκε τελικά ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων εκτόπισε την παραγωγή τροφίμων. Θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ των δύο. Τα βιοκαύσιμα ως εναλλακτικός τρόπος ε, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Γιατί έχουμε συγκεκριμένου ε, ενεργειακού στόχου και στόχου για τι κλιματικέ αλλαγέ που θα πρέπει να λάβει υπόψη και τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και τα βιοκαύσιμα. Και αν δεν κάνουμε μια διαφοροποίηση και ένα άνοιγμα προ αυτού του τομεί, δεν πρόκειται να εγγυηθούμε την ενεργειακή μα ασφάλεια, που είναι εξίσου σημαντικό θέμα με την επισητιστική μα ασφάλεια. Γι' αυτό και ο πρόεδρο Γιούγκερ μου ζήτησε να έχω σχέσεις και να ενημερώνω όχι μόνο έναν αντιπρόεδρο, αλλά δύο. Τον κύριο Κατάινεν για τα οικονομικά θέματα, τις οικονομικές δραστηριότητες και την Σλοβένα αντιπρόεδρο, την κυρία Μπράτουσεκ, που είναι αρμόδια για θέματα ενέργειας, γιατί η ενέργεια και τα τρόφιμα είναι αλληλένδετα ζητήματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια οριζόντια συζήτηση για να για να υλοποιήσουμε ταυτόχρονα το στόχο της επισητιστικής ασφάλειας αλλά και της ενεργειακής μας ασφάλειας. Ευχαριστώ.